Συναδελφοί, αν μπορούμε να ακούσουμε να καταρχάσουμε τις αποφάσεις των συντονιστών που συνεδρίασαν νωρίτερα. Το σχέδιο μίας διάτηξης έγινε δεκτό. Εν συνεχεία το πρώτο θέμα για την μαύρη λίστα των αερομεταφορέων. Ε, όλες οι πληροφορίες δόθηκαν τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και εάν δεν υπάρχουν σχόλια για αυτή τη μαύρη λίστα σε πέντε μέρες θα γράψει ο Πρόεδρος μια επιστολή στον Επίτροπο Κάλλας. Με συνεχεία είχαμε μια ε, απόφαση για την επιτροπολογία των likes και ακούσαμε όλες τις προφορίες από την Επιτροπή. Ο Επίτροπος Κάλλος μας έκανε μία ενημέρωση στις 29 Οκτωβρίου από το Συμβούλιο όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους και ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, εκ μέρους της Επιτροπής θα υποβάλουμε ένα υπόμνημα για απόρριψη και θα δούμε τι θα υποβληθεί και από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Όσον αφορά τους εισηγητές, επιλογή εισηγητών, η πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την συμφωνία οχημάτων στις διεθνές μεταφορές στα πλαίσια του ΟΗΕ και της αρμόδιας επιτροπής ζητήσαμε από την κυρία Τίκαρτ να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας σε συνδυασμό με την έκθεση για τους ταχογράφους, για τις ε, γνωμοδοτήσεις. Η απόφαση των συντονιστών για τις περισσότερες ήταν να μην αναλάβουμε δράση, να μην κάνουμε τίποτα. Η απόφαση για το GNSS με την Ουκρανία, η γνωμοδότηση, η ανακοίνωση για την ενιαία αγορά, το κανονισμό του Συμβουλίου που καθιερώνει ένα σύστημα μεταφοράς ε, ραδιενεργού υλικού, την πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 7098 για τα καύσιμα πετρελαίου και ντίζελ. Εδώ θα ορίσουμε ε, εισηγητή για την γνωμοδότηση βάσει του κυκλικού συστήματος του συστήματος εναλλαγής. Ε, όλα τα άλλα, η αναφορά στο Συμβούλιο για τη φορολόγηση, για την προμήθεια αγαθο, προμήθειες αεροπλάνα, πλοία, φοδιασμούς κλπ. Και επίσης όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, σε σχέση, μαζί με την επιτοπή του ΟΗΕ για τα οικονομικά ζητήματα και την έκθεση για την Επιτροπή που υλοποιεί τη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και την ETF. Ανακοίνωση για τα αυτοκίνητα, 20 πρόγραμμα δράσης, το αναβάλαμε αυτό για αργότερα όταν η Ήτρε θα έχει εκδώσει την έκθεση της. Δεν θα κάνουμε επίσης τίποτα για την συνεργασία καινοτομιών, και επίσης για το Ταμείο Συνεχής Ετήσια Έκθεση, επίσης εκεί δεν αναλαμβάνουμε γνωμοδότηση. Ε, όσον αφορά την, το νομοθετικό πλαίσιο και τα, τα ναυτιλιακά απορρίμματα, ο κύριος Δανέλης ε, θα αναλάβει τη γνωμοδότηση αυτή μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ναυτιλίας και Τουρισμού. Επίσης για την ε, διεύρυνση, για την χρηματοδότηση της Κροατίας. Για την προετοιμασία προς δεν θα αναλάβουμε γνωμοδότηση. Επίσης για την εσωτερική αγορά και τη βαθμολόγηση, επιτροπολογία, ε, υπόψη τα, τα φυλάδια 25-26, ενημερωτικά φυλάδια 25-26 για το ETS είχαμε μια νέα πρόταση από τον αρμόδιο επίτροπο περιβάλλοντος να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία σε, κοινή επιτροπή υπό τον κανόνα 51 για ε, από την ΙΜΚΟ διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς εγκρίθηκε από τους προέδρους και για την ε, φορολόγηση των σιδηροδρόμων στη Γαλλία. Ο πρόεδρος θα γράψει τον Επίτροπο Κάλλας για να μας διευκρινίσει αν αυτή η πολιτική είναι ένομη. Τώρα, σαφήνεια όσον αφορά τις επιτρεπόμενες αποσκευές των επιβατών, αεροπλάνων λέει, σε αεροπλάνα, ε, αυτό δεν θα κάνουμε τίποτα αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση όσον αφορά την απόφαση για την τροποποιημένη οδηγία 126 του 2000 για μια κάρτα οδηγών και επίσης οι διαβουλεύσεις για τους ταχογράφους υπό την Κυπριακή Προεδρία θα συζητηθούν με, υπό την παρουσία του Αντιπροέδρου Κικάλ. Επίσης, ζητούμε μία συνάντηση με όλους τους ηγητές στην αρχή του νέου χρόνου και η θέση του κυρίου Ρίκαλ είναι να ζητήσει διευκρινήσεις για την απόφαση που ελήφθη από την ΑΦΚΟ. Υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις για τις αποφάσεις αυτές. Εάν όχι, τότε γίνονται δεκτές και σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους εναπομείνοντες συντονιστές των ε, ΔΕΔ, Ευρωπαϊκών, ε, Ευρωπαϊκών Δικτύων, τον κύριο Balance, Brinkhorst, Σέτσι, Σάβαρη και Κόξ. 10 λεπτά. Α, ναι, εδώ. 10 λεπτά για τις ε, εισηγήσει τους. Είναι λίγο σύντομος ο χρόνος, αλλά περισσότερα θέματα μείναν εκρεμή από ότι αυτά που ξεκινήσαμε, οπότε παρακαλώ αν μπορείτε να είστε ε, σύντομοι και ε, τα μέλη παρακαλώ επίσης να είναι σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κυρίες και κύριοι, θα σας αναφέρω για το πρόγραμμα προτεραιότητας αριθμό 17 που αποτελεί μια κεντρική σύνδεση από Ανατολή μέχρι Δύση μεταξύ του, και της του Παρισιού και της Μπρατισλάβας διερχόμενο από μια άλλη πρωτεύουσα, τη Βιέννη καθώς και περιφερειακές πρωτεύουσες όπως μόνο το Τουγάρδι και πρωτεύουσες διαφορών Λέντερ μεταξύ άλλων και το Στρασβούργο επίσης. Η πρόοδος υπήρξε εντυπωσιακή. Είχα το προνόμιο να παρακολουθώ αυτό το φάκελο από την αρχή όταν επιλέξαν τα πρώτα πέντε έργα προτεραιότητας χωρίς διακοπή από μέρους μου και μπορώ να σας αναφέρω ότι σήμερα οι τελευταίες στατιστικές που ετοιμάσαμε αναφέρουν ότι το 43% της όλης γραμμής βρίσκεται ήδη σε λειτουργία θα χρειαστεί να επαναυπολογίσουμε αυτό το ποσοστό, διότι πριν από λίγες μέρες, στις 23 Νοεμβρίου, εγώ παρευρέθηκα μαζί με πολλούς άλλους στην, ε, στα εγγένεια στις ε, σύνδεσης ε, μεταξύ Βιέννας και Σάλτσπορ και είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι με, και Πόλτεν, συγγνώμη, με ε, πολλές σύραγγες και θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της όλης γραμμής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η γραμμή έχει κοστίσει μέχρι τώρα 680 εκατομμύρια ευρώ. Τα 600 προήλθαν από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και τα υπόλοιπα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει το Ταμείο Συνοχής που στην περίπτωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας έπαιξε σημαντικό πρόσθετο ρόλο. Ε, Ένα από τους κύριους ε, στόχους μας ήταν πάντα η διατροπικότητα. Σημαντικά αεροδρόμια και ε, υδάτινες διαδρομές και υπάρχουν κάποια εξαιρετικά παραδείγματα. Το αεροδρόμιο Σάλντεγκόλ του Παρισιού έχει διεθνή σύνδεση. Στη Βιέννη ο νέος κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός που βρίσκεται υπό κατασκευή θα συνδέεται απευθείας με τις αερομεταφορές και αναζητάμε μια καλή λύση για την πόλη της Στουτγάρδης και του Μονάχου. Ενθαρρύνουμε ωστόσο να το βρουν και για τον προγραμματισμό έχουμε, μπορούμε να προσφέρουμε εμείς το 50% της χρηματοδότησης ε, του προγραμματισμού αυτών των έργων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τις προσπάθειες της Γαλλίας και της Αυστρίας. Αυτές οι δύο χώρες ε, δουλεύουν επισταμένα για την ανάπτυξη των γραμμών ε, στα εδάφη του και τι συνδέσει με του γείτονε. Υπήρξαν κάποιε δυσκολίε στη Γερμανία, ειδικότερα τα διασυνοριακά τμήματα προ Γαλλία και Αυστρία. Και στη Σλοβακία οι προγραμματισμένε ε, συνδέσει βρίσκονται υπό επανεξέταση. Συζητήσαμε λεπτομερώς όλα αυτά τα προβλήματα στην εκθεσή μου θα βρείτε τις δραστηριότητες από τα μέσα του περασμένου χρόνου στην προηγούμενη μου έκθεση, πάντα και διαβάζω την προηγούμενη μου έκθεση, όταν έρχομαι να συναντήσω την Επιτροπή Μεταφορώ, εκεί είχα επισημάνει τα σημαντικότερα βήματα για την επόμενη περίοδο και τώρα κλείνουμε αυτή την επόμενη περίοδο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας αναφέρω ότι Αυτά τα μέτρα υλοποίησης υλοποιήθηκαν. Πρώτα απ' όλα το δημοψήφισμα στη Στουτγάρδη ε, αποτελούσε μείζον ζήτημα το Νοέμβριο του 2011. Αυτό το δημοψήφισμα έλαβε χώρα και το ε, πρόγραμμα Stuttgart 21 θα μπορέσει να ακολουθηθεί, να συνεχιστεί και οι εργασίες ξεκίνησαν ξανά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο τμήμα στο καρδιούν που είναι το πιο περίπλοκο και το πιο ακριβό ε, τμήμα της γραμμής ε, σύνδεσης με την Πρατισλάβα. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης αναβλήθηκε λίγο μέχρι τα τέλη του 2020, αλλά οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά. Η άλλη προτίμηση, μάλλον επιθυμία, ήταν το άνοιγμα της γραμμής Μονάχου Augsburg που επιτρέπει ύψηλε ταχύτητε και που έχει υλοποιηθεί μέχρι το Δεκεμβρίου, υλοποιήθηκε μέχρι τέλη του Δεκεμβρίου πέρυσι. Η μετάβαση έγινε κατά το χειμερινό, ε, τα χειμερινά δρομολόγια. Το νέο ΤΖΒ από το ε, Μασαλίας ε, ε Μα ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η σύνδεση και τέλος ξεκίνησαν οι εργασίες του... σε προγραμμένες γραμμή Clearing Saife στη Βιέννα που επιτρέπει τη σύνδεση με το αερο... του αεροδρομίου με άλλες ε, πόλεις μαζί με την κατασκευή του νέου συντηροδρομικού σταθμού. Ξεκίνησαν οι εργασίες τον Απρίλιο φέτος. Ανέφερα το Σάλτσπορ και τη Βιέννη και άλλα έργα βρίσκονται υπό εξέταση. Έχω την αίσθηση ότι μετά από την τελευταία μου επίσκεψη στην Πρατισλάβα ότι προοδεύουμε αλλάζοντας την αρχική ιδέα του σύραγγας ε, του Δούναβη σε μια άλλη λύση η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού καθώς και η ανατολική σύνδεση του αεροδρομίου της Βιέννης ε, θα αλλάξει, η οποία θα απαιτήσει επικοδομητική και φιλική συμφωνία μεταξύ των τριών γειτονικών χωρών που συνορεύουν σε εκείνο το σημείο, Αυστρία, Σλοβακία και Ουγγαρία. Αλλά και αυτές ενθαρρύνθηκαν από την Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα το μέλλον, πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ε, καταργήσουμε έτσι τα σύνορα, θα εφαρμόσουμε τις ε, ε, συνδυασμένες μεταφορές. Κάθε κράτος μέλος αισθάνεται την ευθύνη, διότι πρέπει να συνεργαστούν με τους γειτονές τους για την ε, οικοδόμηση των δικτύων μεταφορών και φυσικά ανυπομονούμε να δούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τι στο πλαίσιο αυτού θα επιτραπεί στην Επιτροπή να ξεκινήσει και τι θα μπορέσει η Κομισιόν, πώς θα μπορέσει η Κομισιόν να ενθαρρύνει τα κρατημέλη να κάνουν τι. Γνωρίζουμε καλά ότι στο νέο μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις. Τουλάχιστον έτσι έχουν προταθεί από την Κομισιόν. Και η γραμμή που σας παρουσιάζω εγώ αυτή τη στιγμή θα προσθεθεί σε δύο μεγαλύτερα έργα. Το νέο διάδρομο Στρασβούργου-Δουναβή από το Στρασβούργο μέχρι το Σούλινα στην ε, Μαύρη Θάλασσα με ένα κλάδο που θα ακολουθεί το σημερινό PP17 στο τιαρδι Μόναχο και το άλλο μέσω Φραγκφούρτης Νιρεμβέργης και Ρέγγενσμπουργκ. Θα ακολουθεί δηλαδή τον Μάιν και τον Δουναβή που αυτή τη στιγμή έχει τον αριθμό PP80. Ε, έτσι θα φτάνουν στη Βιέννη και το πιο μικρό κομμάτι του σημερινού PP17, e το δυτικό κομμάτι, ε, Παρίσι με Στρασβούργο, θα αποτελέσει κομμάτι του διαδρόμου Λισαβόνα-Στρασβούργου. Θα συναντώνται κοντά στα κεντρικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και θα ανοίγουν το δρόμο προς δύο κατευθύνσεις την Ευρώπη. Και φυσικά η διαδρομή αυτή θα είναι ε, πολυτροπική. Θα, με το PP17 προσπαθούμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι διάφοροι τρόποι μεταφορών. Ε, παρουσιάσαμε τις προάλλες ε, στο πλαίσιο μιας ημερίδας τις καλύτερες συνδέσεις που μπορούμε να επιτύχουμε με σιδηρόδρομο και αεροπορικό. Έχω ολοκληρώσει κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάλαντς. Ευχαριστώ κύριε στον κατάλογο έχω τους κυρίους Gross, Χέρτουγκ, Κράμερ, Βίλ Λίχτεμπεργκερ και την κυρία Μάισνερ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Μάθιο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συντονιστή για την έκθεσή του είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή την οποία έπρεπε να επεξεργαστείτε ως ε, συντονιστής και σε έχω τρία ερωτήματα που βασίζονται στην εμπειρία σας. Και ως, αν δεν είσαι Γερμανός έχεις ακούσει για το θέμα της Τουτγάρδης και θα ήθελα να ακούσω από εσά τι μας συμβουλεύετε ως μέλη του Κοινοβουλίου. Ή πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις ή να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Όταν τέτοια έργα στραβώνουν. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερο ερώτημα. Σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτό το μήκος, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε στο Κοινοβούλιο ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο επικεντρώνεται, α, το οποίο βασίζεται ιδιαίτερα στο Συμβούλιο, διότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν κατά πολύ συμφωνήσει ότι το έργο αυτό είναι σωστό, είναι καλό, αλλά πρέπει να πείσουμε τα κράτη. Αυτό το έργο το οποίο διαπερνά αρκετές χώρες, πολλαπλές χώρες, δεν είναι εξαιρετικά κατάλληλο για να υποστηρίξει και να εδραιώσει αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, θα θέλουμε την άποψή σας. Το τρίτο, ε, τρίτη ερώτηση, μιλάμε για νέα έργα, νέα χρηματοδοτικά μέσα. Τα θεωρείτε επαρκή ή πιστεύετε ότι χρειάζονται και περαιτέρω βήματα, περαιτέρω μέσα για να μπορούν να σταθεροποιήσουν μακροπρόθεσμα αυτά τα καινούργια έργα. Ο κύριος Έρτογκ. Ευχαριστώ κύριε Μπάλας για την παρουσίαση, εισήγησή σας και την τελευταία φορά μας είχατε εντυπωσιάσει αναφερόμενο σε όλες τις εξελίξεις, σε, όλα, σε όλη την πρόοδο. Θα ήθελα κύριε Μπάλλας να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε τώρα τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχουμε τη νέα ατζέντα και έχουμε αυτά τα 30 έργα προτεραιότητος σε, σε συγκεκριμένους διαδρόμους, τα οποία έχουμε ενσωματώσει, εκτός από μερικές λίγες εξαιρέσεις τι οι, αυτές οι εξελίξεις τώρα οι σημερινές συνάδουν με αυτούς τους διαδρόμους που έχουμε αποφασίσει διότι έχετε πλέον κάποια εμπειρία στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τα διάφορα κράτη-μέλη και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη θέση σας και αυτή και στις διαβουλεύσεις που θα κάνουμε με τα άλλα μέρη. Η κυρία Μάισνερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις ερωτήσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε στη Σλοβακία και είπατε ότι είναι υποσκέψη. Τι σημαίνει αυτό. Είναι θετική προσέγγιση ότι θα γίνει οριστικό ή είναι αβέβαιο, μέλλον και αβέβαιο. Διότι για τα διευρωπαϊκά μεταφορών ε, ε, θέλουμε να αποφύγουμε έργα τα οποία ξεκινάνε αλλά δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Ε, Έχουν να παίξουν ρόλο λοιπόν και τα κράτη-μέλη. Δεύτερη ερώτηση έχουν σημειωθεί με κόκκινα έργα τα οποία θα αρχίσουν μετά το 2013. 2013. Όλοι ξέρουμε, ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να μειώσουν τη διασύνδεση και η Επίτροπος ο Επίτροπος ε, θέλει να προχωρήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία αφορούν τη Γερμανία και την Αυστρία και τι θα γίνει α, εάν αυτά τα χρήματα, οι πιστώσεις δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν. Ο κύριος Κράμερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ για την παρουσίασή σας, σας έχουμε ακούσει επανειλημμένος. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί για τη Στουτγάρδη, δηλαδή όλα έχουν αποφασιστεί εκτός από τα χρήματα. Ακριβένουν συνέχεια οι δαπάνες, τι θα γίνει με αυτό το τούνελ, αλλά το βασικό σημείο είναι η νέα διαδρομή Στουτγκάρδης Ούλμ, η οποία θα γίνει επειδή ο παλαιός άξονας δεν ενδείχνει πλέον για τη μεταφορά αγαθών. Ξέρουμε ότι όσοι φτάνουν στη Στουτγάρδη μόνο το 30% πηγαίνει περαιτέρω στην Ούλμ για τρία δισεκατομμύρια τώρα χτίζεται ένας καινούριος ε, άξονας, ο οποίος έχει την ίδια κλίση, είναι το ίδιο απότομος, ε, για μια, ένα πολύ μικρό ποσοστό μεταφορών αγαθών που πηγαίνει στον τελικό προορισμό. Τώρα, εάν μεταφορές αγαθών πηγαίνουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον παλιό ή τον καινούριο άξονα, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι προστιθέμενη αξία σε αυτό το νέο έργο. Γιατί χρηματοδοτείται αυτή η νέα, ο νέος άξονας, παρόλο που έχει σαφώς μειονεκτήματα είναι η προσέγγιση για όλα τα νέα έργα, για νέες ε, διαδρομές, για νέες επεκτάσεις η ίδια, είναι η ίδια προσέγγιση ή, περιορι... ή εξειδικεύεται ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε έργου. Η, κυρία... Geislinger Steiger, hätte ich auch angesprochen. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω μετά την ερώτηση του κ. Κράμερ για τις μεταφορές αγαθών. Έχω όμως και κάτι άλλο το οποίο με ανησυχεί. Λέγεται ότι η εργασία στη Στουτγάρδη, στο συνδρομικό σταθμό, θα καταβληθούν από την UTNT. Δηλαδή, δεν θα υπάρξουν νέες πιστώσεις για τον σταθμό στη Στουτγάρδη, αλλά θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα κεφάλαια. Σωστό ή λάθος. Ο πρόεδρος. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, ευχαριστώ. Και εγώ για τον ομιλητή. Ξέρω και εγώ τα πλεονεκτήματα της επέκτασης, της βελτιώσεις που γίνονται για να μειωθεί ο χρόνος και να βελτιστοποιηθούν οι γραμμές. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να έχουμε θετικά σημάδια στις μεταφορές αγαθών που θα ήταν, δηλαδή στην αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών. Δυστυχώς. Τώρα, μεταξύ Γαλλίας-Γερμανίας, όσον αφορά τις ιδιασμένες μεταφορές ε, στην ε, μεταφορές ατόμων, ε, επιβατών. Ε, ακούω ότι κάτι τρέχει, αλλά τι πληροφορίες έχετε εσείς. Τώρα, όσον αφορά το τρίγωνο αυτό στο Brockhausen, θα διασυνδεθεί. Βέβαια, οι συνδρομικές μεταφορές, οι πραγματικές μεταφορές είναι πιο, βέβαιες, πιο σίγουρες, πιο ασφαλείς από ότι στο αδικά δίκτυα. Αλλά αυτή η διασύνδεση και αυτή η διακλάδωση προς το Milhausen-Brockhausen, αυτό το τρίγωνο δηλαδή, δεν προχωράει όσο θα έπρεπε. Υπάρχει καθυστέρηση σε αυτή τη διακλάδωση. Ε, και κάτι άλλο στον, ε, για την Πρατισλάβα, σε αυτό το θέμα. Από ό,τι ξέρω, τα προβλήματα δημιουργούνται επειδή απερίφθη μία αίτηση η οποία έχει υποβληθεί και γι' αυτό δεν επιλέχθηκε η καλύτερη λύση. Δεν, επιλέχθη, δεν μπορούσε να επιλεχθεί η καλύτερη διαδρομή διότι απερίφθη το αίτημα κατασκευής. Τώρα, το να συνδεθεί και το αεροδρόμιο σε αυτή τη γραμμή δεν είχε προβλεφθεί αρχικά με τη διασύνδεση των δύο συνδρομικών σταθμών. Καλά, αυτό είναι το ελάχιστο αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτό το κόλλημα που έχει σημειωθεί στην Πρατισλάβα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παλζάς, αν μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ. Στουτγάρδη 21. Τι μάθαμε από αυτή την περίπτωση και από την Κομισιόν, από πλευράς Κομισιόν. Ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα καταρχάς. Πρώτον για την πόλη και δεύτερον για το κρατήριο της Βάδης Βιτεβέργης. Και βεβαίως εν συνεχεία σε όλη την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Για μένα το ζουμί, το ζουμί της ιστορίας είναι ότι μια πολιτική στήριξη δεν διαρκεί για πάντα. Στην αρχή υπήρχε μια βούληση, υπήρχε μια σύμπνοια, μια υποστήριξη. Ας το πούμε ότι δεν υπήρχε αντίρρηση, δικαιολογημένη αντίρρηση ή αντίσταση σε αυτό το έργο. Με τον κύριο Κράμερ πριν από 7 χρόνια είχαμε διαφορές απόψεων, αλλά μετά είπαμε ότι η απόφαση ανήκει στον Τεμπλάντε και στην πόλη και ας δούμε τι θα αποφασίσουν αυτοί ένταξη άλλαξη κατάσταση και οι σχέσεις ε, του, του, του, του, πληθυσμού των πολιτών στην κυβέρνηση κλπ. Ε, αυτά τα μακροπρόθεσμα έργα άπτονται πολλών κυβερνήσεων, όχι μόνο στο κράτος μέλος, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη, στις διάφορες ε, χώρες οι οποίες, οι οποίες ε, ε, επηρεάζονται από αυτά τα έργα. Παραδείγματο χάρη πολλές φορές για ένα έργο έχω μιλήσει με πέντε υπουργού από το 2005. Αλλάζει δηλαδή και η κυβέρνηση η αρμόδη και οι απόψεις. Το θέμα είναι εάν το έργο αυτό έχει γίνει πολύ πιο ακριβό. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, διότι στη φάση προγραμματισμού οι δαπάνε δεν είναι τόσο μεγάλε. Στην συνεχεία βεβαίω διαπιστώνεται ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα ε, και τελικά ξεπεράστηκε ένα κατόφλι. Εν συνεχεία σημειώθηκε μια αντίδραση, άλλαξε η κυβέρνηση και η εμπειρία μου ήταν ότι Εάν υπάρξει μια πολιτική στήριξη πρέπει κανείς να προσπαθήσει να τη διατηρήσει. Πρέπει με κάθε αλλαγή κυβέρνησης, ε, ίσως και κάθε χρόνο. Πρέπει κανείς να επανέρχεται στα ίδια ερωτήματα για να εξασφαλίσει τη στήριξη. Παραδείγματο χάρη η στήριξη για, τις ε, κίνηση, για την κίνηση που λέγεται στα γερμανικά Magistrale für Europa. Äh, äh, Είναι μια κίνηση πολιτών η οποία ε, αρχίζει και διευρύνεται και ενδιαφέρει όλο και περισσότερους. Και σε αυτή η κίνηση στηρίζει τους σιδηροδρόμους. Το TGV, το TGV, ε, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές από τη Γαλλία στη Γερμανία και αντίστροφα. Και είναι πολύ δημοφιλή αυτές οι ταχείες συνδρομικές γραμμές. Και, και δουλεύουν και πολύ καλά. Ο συνάδελφός μου, κύριος Βίνγκ, μπορεί να μιλά για όλα τα προσόντα των συνδυασμένων μεταφορών. Το έκανε και, και χτες. Είναι γεγονός ε, ότι και οι άλλες γειτονικέ χώρες έχουν τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη πώς μπορούν συνδυασμένα να εκπονήσουν ένα χρονοδιάγραμμα. Ε, αν ε, έχει κανείς εκατοντάδες τρένα τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες γραμμές, κάθε μέρα ε, ένα συνδυασμό ε, προσπαθειών ε, είναι πολύ σημαντικός. Επίσης είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα του τριγώνου, στην, του χημικού τριγώνου στην Νότια Γερμανία. Η χημική βιομηχανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να βγουν τα προϊόντα προς τα έξω, εξαγωγές, και αυτή είναι η καλύτερη λύση, το λεγόμενο χημικό τρίγωνο. Ε, αφορά προϊόντα τα οποία έχουν χημικά προϊόντα, ουσίες χημικές, ε, χαμηλής αξίας. Και όλες οι ενδείξεις μας ε, λένε ότι αυτά τα δίκτυα πρέπει να επεκταθούν παρόλο που εγώ πιστεύω ότι το το πλαίσιο δεν επαρκεί, αλλά η αρχική πρόταση της Κομισιόν για τα 15 δις ήταν σωστή και σε συνεργασία με το Ταμείο Συνοχής βεβαίως. Ε, ήταν εφικτό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η πολιτική μεταφορών. Κάθε περικοπή είναι επικίνδυνη και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Η διευκόλυνση για την Ευρώπη. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, αυτού του έργου, διευκόλυνση για την Ευρώπη. Έχω ασχοληθεί και με την πολιτική συνοχή και αυτός ο μηχανισμός εξελίσσεται από τη βάση, από τα κάτω προς τα πάνω. Όταν λοιπόν προσιαστούν οι διάφορες προτάσεις, πρόκειται μάλλον για μικρά έργα, από τα κράτη, από τις κυβερνήσεις, δημιουργείται ένα μοσαϊκό με όλα αυτά τα συστατικά στοιχεία και όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά ή θεωρούνται σημαντικά για αυτούς που τα επεξεργάστηκαν. Αλλά μία αληθινή προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να την εντοπίσουμε με τη μέθοδο την οποία έχει χρησιμοποιήσει η Κομισιόν στο CEF. Εάν δούμε δηλαδή τα μεταφορικά ρεύματα πέραν των συνόρων, εν συνεχεία να τα δούμε τις ροές αυτές τα σύνορα, τις διασυνοριακές μεταφορές, και τις συνδυασμένες μεταφορές. Άμα εξετάσετε με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο, τότε θα δείτε ότι πραγματικά λειτουργεί. Ταυτόχρονα η Κομισιόν πολύ προσεκτικά συζήτησε με τα κράτη-μέλη για να τα πείσει για τα πλεονεκτήματα. Αλλά εάν εξετάσει κανείς την κατάσταση από το υψηλότερο επίπεδο, θα δει κανείς ότι εκεί είναι πολύ καλύτερος ο προγραμματισμός. Τώρα, είναι είναι είναι οι είναι οι διάδρομοι. Αυτή ήταν μία προϋπόθεση της προετοιμασίας και μία πάρα πολύ σύγχρονη προσέγγιση των ευρωπαϊκών μεταφορών. Αυτό είναι ένα στοιχείο του ανταγωνισμού μας. Εάν είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ολόκληρη η Ευρώπη μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Το αποτέλεσμα όλων των ε, διαβουλεύσεων ήταν το διευκόλυνση για την Ευρώπη. Στη Σλοβακία συζητήσαμε το τούνελ κάτω από το ποτάμι. Α, ονειρευόταν μάλλον ένα τούνελ κάτω από το ποτάμι. Το συζητήσαμε, είναι ένα δαπανηρό έργο και μετά από πολλές αναλλαγές κυβερνήσεων η ιδέα αυτή άλλαξε. Αρχές Σεπτεμβρίου ήμουνα στην Πρατισλάβα, μίλησα με τον κύριο Κοτσάτεκ, τον Υπουργό Μεταφορών. Είναι νέος στον, καινούργιος στον τομέα των μεταφορών, όχι νέος, νέο μέλος της κυβέρνησης. Κατανοεί το θέμα και είχε μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση μετά από την επίσκεψή μου ακούσαμε την καλή είδηση ότι η κυβέρνηση έχει πλέον κατά κάποιο τρόπο εγκαταλείψει αυτή την ιδέα και θα παρουσιάσει νέες ιδέες. Αυτή είναι καλή είδηση. Η Μπρατισλάβα έχει μικρό αεροδρόμιο, η Βιέννη έχει ένα μεγάλο αεροδρόμιο, τα δύο αυτά αεροδρόμια είναι πολύ κοντά και θα μπορούσαν θαυμάσια να αλληλοσυμπληρώνονται. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή και ταχεία ε, σύνδεση των δύο αεροδρομίων. Αυτό είναι εφικτό. Ε, και μάλιστα συνεχώς αναφέρεται ότι παλιά επί Κάις επί αυτοκρατορίας υπήρχε το τραμ, το περίφημο τραμ που συνέδε την Πρατισλάβα με τη Βιέννη. Δεν μιλάμε γι' αυτό βεβαίως τώρα. Ε, κύριε Κράμα, ως συνήθως μου θέτει... Ε, ναι, λίγο πιο υπερταχεία λέει ο πρόεδρος παρακαλώ. Συντομεύεται. Λοιπόν, ε, σημείωσα την ερώτηση του κυρίου Κράμερ, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θα κοιτάξω να, να δω τι συμβαίνει. Όλη αυτή η γραμμή δεν λειτουργεί χωρίς την Στουτγάρδη και για τους επιβάτες και για τα εμπορεύματα. Και τα δύο πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ έχω κάνει αυτή τη διαδρομή πολλές φορές, ξέρω τα γεωγραφικά δεδομένα και θα επανέλθω να σας απαντήσω. Αν με επιτρέπετε. Το ίδιο επίσης για τις εργασίες των γραμμών στη Στουτγάρδη. Δεν ξέρω, επί των γραμμών, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολλά πράγματα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εμείς κατασκευάζουμε γραμμές, χρειαζόμαστε συνεχώς βοήθεια για την κατασκευή νέων, επέκταση των γραμμών και αυτά τα έργα ανήκουν στους Δήμους ή στον Οργανισμό Γερμανικών Σιδηροδρόμων, στην Deutsche Bahn. Θα σας απαντήσω όμως. Για το... Θα σας απαντήσω την ερώτησή σας. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Μπρίνκχορτ, να καλωσορίσω 14 φοιτητέ από την École ε, Nationale de la Sécurité de la Mer. Νομίζω ότι είναι ε, για την αυτιλή αυτό όλο που διάβασα στα αγγλικά. Τους καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συνεδρίαση σήμερα. Συνοδεύεται ε, από τον διευθυντή τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους φοιτητέ, οι οποίοι είναι φοιτητέ σε ναυτιλιακά θέματα. Κύριε Μπρίγχορστ, νομίζω ότι ήρθε η σειρά σας. Ε, πρόγραμμα προτεραιότητας 6, Λιόν, Τεργέστη, Κόπερ, Λουμπλιάνα, Βουδαπέστη και Ουκρανία φτάνουμε και μέχρι το Πεκίνο ή όχι. Δέκα λεπτά λοιπόν για την παρουσίασή σας. Θα σας ήμουν ευγνώμων να τηρήσετε και το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάντα να έχουμε εδώ στην Επιτροπή σας ε, και να σας κάνω έναν απαλλαγισμό των όσων συνέβησαν πέρσι θα έχετε λάβει, ε, ή τουλάχιστον εγώ σας την έστειλα, την ετήσια έκθεση. Να περάσω λοιπόν σε κάποιες πιο πρακτικές και ίσως και πολιτικής φύσεως ε, παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ότι παρά το πολύ δύσκολο πολιτικό κλίμα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ε, για τις περαιτέρω προσπάθειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μια κάποια πρόοδο για ένα από τα βασικά ε, στοιχεία του διαδρόμου της ε, Ανατολικής Δυτικής Ευρώπης. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για τα βασικά σημεία. Το βασικό βεβαίως είναι το διασυνοριακό τμήμα ε, Λιών Τωρίνο μεταξύ Γαλλίας και ε, ε, ε, Ιταλίας και το δεύτερο τμήμα είναι το Τεριέστη Ιντιβάτζα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας και φυσικά υπάρχουν και κάποια νεότερα για την Ουγγαρία και τη Σλοβενία που είναι πρόσφατα στοιχεία αλλά καταδεικνύουν ότι η πολιτική βούληση στις τέσσερις βασικές χώρες της νότιας γραμμής υπάρχει παρά τις αντικσοότητες. Κυρίως μας ενδιαφέρει η γραμμή Λιών Τωρίνο Εκεί υπεγράφει μια νέα συμφωνία μεταξύ των αρχών Γαλλίας και Ιταλίας. Μετά την άφηξη του Πρόεδρου Μόντε, ε, Μόντι, ο, ο νέος Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ιταλίας ε, να ε, συνεχίσει την διαδρομή αυτή. Υπήρξε λοιπόν μια συνεννόηση και η συμφωνία αυτή αποτελεί πλέον το θεμέλιο προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα από τη φάση της μελέτης ε, στο, σχέδιο, στο στάδιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής. Τι αποφασίστηκε. Καταρχάς, ε, νέα κατανομή του κόστους που είναι πολύ σημαντικό υπήρχε και το θέμα της νέας χάραξης της γραμμής ε, και την εφαρμογή σε δύο στάδια, αλλά και νέα διαδικασία διακυβέρνησης. Και θα γίνει και η κύρωση, φαντάζομαι, ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα μετά από την σύνοδο της επόμενης εβδομάδας, Μόντι ε, Ολάντ, ε, και ελπίζω να υπάρχει και μια νέα συμφωνία, διότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του προγράμματος, κάτι το οποίο είναι καινοτόμο αυτό καθε αυτό και φαντάζομαι ότι θα ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχε τέτοιε πρωτοβουλίε τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τι ακριβώ έχει γίνει από πλευρά έργων. Υπάρχει η προετοιμασία τη σύραγγα τη Μανταλένα, που όπω ξέρετε έχει καθυστερήσει παρά τι πάρα πολλέ δυσκολίε. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει και έχουν ξεκινήσει και ανασκαφέ για το ιταλικό τμήμα τη σύραγγα. Ε, θα ξεκινήσουν σύντομα. Μιλάω βέβαια ε, εδώ υπό την εποπτεία τη συνεργάτη μου η οποία θα σα δώσει και τι ημερομηνίε. Από πλευράς Γαλλίας, ε, τα επόμενα έργα τα οποία θα γίνουν είναι η παράταση ε, ε, του σύραγγα του Σαμαρτάν που έχει πρόσβαση και στο λιμάνι και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει και τμήμα της βασικής σύραγγα. Υπάρχει επίσης και μια ιστορική γραμμή εδώ μεταξύ Λιών και του Τωρίνου. Ανέκαθεν υπήρχαν πιέσεις, ανέκαθεν ενδιαφερόταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπήρχαν και προθεσμίες για να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες για αυτή τη νέα γραμμή και έχουν γίνει αρκετά εντατικά όργαν ε, για να βελτιώσουμε το προφίλ της σύραγγας και να εξυγχρονίσουμε και τις εγκαταστάσεις. Αυτά ε, ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2011. Ε, δυστυχώς για τεχνικούς και διοικητικούς λόγους ε, η, τα εγκαίνια αυτού του ιστορικού τούνελ καθυστέρησαν αλλά με χαρά μπορώ να σας πω ότι η σύραγγα αυτή πλέον έχει ξανανοίξει, είναι διπλής κυκλοφορίας και χρειάστηκαν πιέσεις και σε υψηλό επίπεδο ε, διαχείρισης και από πλευράς Ιταλίας και από πλευράς Γαλλίας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, διπλή κυκλοφορία σύραγγα σε πλήρη λειτουργία. Και ελπίζουμε ε, ότι θα ξεκινήσει, έχει ανοίξει λοιπόν η σύραγγα, αυτή η ιστορική διαδρομή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και φυσικά έχουμε και συνδυασμένες μεταφορές ε, διότι από αρχές Ιουνίου του 2012 έχουν ξεκινήσει και οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι αυτοκινητόδρομοι που μπορούν να μεταφέρουν όλες τις μορφές εμπορευματοκιβώτια μεταξύ Λιών και Τουρίνου. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι είναι και καινοτόμο στοιχείο αλλά δείχνει και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα ε, στοιχεία. Έχουμε τακτικά συναντήσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου και μια πλατφόρμα για τη διαδρομή αυτή, την οποία σύστησα εγώ πριν από δύο χρόνια και μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Δύο λόγια τώρα για τη γραμμή Ιταλία-Σλοβενία. Για ιστορικούς λόγους, η συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας ε, δυστυχώς δεν ήταν πάντα επικοδομητική για ιστορικούς λόγους που οι περισσότεροι από εσά ε, που έχετε ζήσει στην περιοχή ε, συνειδητοποιείτε ποιοι είναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως τώρα το γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων. Και ε, έχουμε μια δομή αντίστοιχη με την γαλλοϊταλική. Τώρα στην Τεργέστη πλέον θα υπάρχει μια ιταλοσλοβενική συνεργασία, μια δομή. Ε, θα υπάρχει ένα ανώτερο αξιωματούχο από πλευρά Ιταλία και ένα από πλευρά Σλοβενία. Και φυσικά ε, θα ξεκινήσουμε από 1η Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχημένοι και θα συνεργαστούν για το προκαταρκτικό σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει εντό ολίγου. Τη διαχείριση του προγράμματος θα την έχει αυτή η κοινή δομή που έχουμε συστήσει και ελπίζω ότι θα είναι και χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρία ε, της γαλλοϊταλικής συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε το τρίτο στοιχείο. Ειλικρινά να σας πω, αν δεν υπάρχει επιτυχία μεταξύ Λιών ε, Τωρίνο, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ε, επιτυχία στα υπόλοιπα. Ε, μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβενίας υπήρχε τεχνική συνεργασία και δεν ήταν και πολύ άσχημη. Εκπήρας όμως ε, να σας πω ότι δεν αρκεί να υπάρχει μόνο τεχνική συνεργασία μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία σε διοικητικό και διευθυντικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που προσπάθησα να κάνω το τελευταίο έτος ήταν να αναπτύσσω τις δύο χώρες, να συστήσουν μια κοινή δομή ε, με βοήθεια σε πολιτικό επίπεδο. Έκανα την πρόταση και στη Βουδαπέστη και στη Λουμπλιάνα, ε, στα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία. Η αντίδραση ήταν θετική εκατέρωθεν και ελπίζω ότι το 2013 θα έχουμε μία επιτροπή και να μπορέσουμε να συστήσουμε μια αντίστοιχη δομή που θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και για να σε υπενθυμίσω λίγο και το πόσο καθυστερημένο είναι αυτό το σύστημα, ακόμα δεν υπάρχει ηλεκτροκίνηση μεταξύ Λουμπλιάνα και, τα, και Ουγγρικών συνέρων. Και αν δεν υπάρξει ηλεκτροδότηση λοιπόν εκεί, πώς θα μπορέσουμε να ε, διασφαλίσουμε ότι θα είναι ομαλή η κίνηση. Επομένω, ε, έχει επιτευχθεί πρόοδος ε, στα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είναι πολύ κοντά στην υλοποίησή τους. Ε, ως συντονιστής βέβαια ε, είμαι κάλλιστα να βοηθήσω να επιταχύνουμε και τα προγράμματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα δυνατό κάτι τέτοιο. Το αρνητικό πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη ε, συνολικά είναι ανασταλτικός παράγοντας και φυσικά οι ε, των δημοσίων οικονομικών ε, δεν βοηθούν καθόλου. Ε, δεν χρειάζεται να σας το πω. Εγώ ήμουν συντονιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια του προϋπολογισμού για το 1997, οπότε κατανοείτε ε, κι εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξο, διότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. ελπίζω λοιπόν στις 3 Δεκεμβρίου να δοθεί το, πρώτο, το πράσινο φως για την γαλλοϊταλική συνεργασία από τους κυρίους ο Ολάντ και Μόντι. Και ε, ολοκληρώνοντα να σα πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται ενεργά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές ε, μεταφορών. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αποκλειστικώ και μόνο στα κράτη-μέλη, ιδίω όταν έχουμε τόσο μεγάλα προγράμματα όπω το Λιόν ε, το Ρήνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ευημερία. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα του χρόνου και να σας πω ότι επετεύχθη κάποια πρόοδος παρά τις αρνητικές ε, στάσεις που έχουν αρκετοί πολλές φορές. Ο κύριος Κανσιάν και η κυρία Λιχτεμπέργεν θέλουν το λόγο. Κάποιος άλλος ο κύριο Καντσιάν καταρχάς. Να υπενθυμίσω στα μέλη όμω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω τις σκέψει σα. Εάν θέλετε το λόγο πρέπει να μου το πείτε. Ο κύριο Καντσιάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρίνκχοστ για το έργο σας και για τη δέσμευσή σας ε, το χρόνο που αφιερώνετε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία ώστε για να μην μιλήσω με όλους τους συντονιστέ, να προσπαθήσω να κάνω τρεις παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και ενδεχομένω θα μπορούσα να λάβω και μία απάντηση για αυτά τα τρία σημεία τους διάφορες ε, συντονιστέ. Ε, καλό είναι να απαντηθούν αυτά πριν από τι εγκρίσεις των διευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών στα μέσα Δεκεμβρίου. Εδώ βρίσκονται και οι συγητές και ο συνάδελφο. Κουμουτσάκος και Έρτοκ που θα πρέπει να σημειώσουν και αυτές τις συναντήσεις. Ε, η ερωτήση είναι η εξής. Σήμερα έχουμε μπροστά μας την έγκριση των συντονιστών για τον συντονισμό για πέρασμα από το modal στο intermodal ώστε να χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές μεταφορών στις διαδρομές προβλέπονται. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό και πρέπει να γίνει αυτή η απλούστευση σε σχέση με τις εμπορευματικές μεταφορές που εγκρίναμε πέρυσι. Αυτός ο συντονισμός λοιπόν θα περάσει από έναν συντονισμό τροπικό και έναν διατροπικό. Ένας δεύτερος προβληματισμός για να καταλάβω κατά την άποψή σας επειδή δεν παρατηρείται επιτάχυνση αυτής της εργασίας και έχουμε μακροχρόνιες προθεσμίες πιστεύετε όλα αυτά εξαρτώνται από τα εδάφη, από τα χρήματα από τι σε τι οφείλεται αυτή η καθυστέρηση η τρίτη σκέψη είναι ότι αν μπλοκάρουμε το διάδρομο σε κάποιο σημείο του μήκους του τελικά θα πάψει να υπάρχει θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τα μπλοκαρίσματα αυτά, διότι θα σημαίνουν το τέλος της εκάστοτε διαδρομής. Η τελευταία μου σκέψη, κύριε Πρόεδρε, τα project bond, τα ομολόγα υλοποίησης προγραμμάτων, ήδη οι πόροι θα χρειαστούν ή θα βοηθούσαν να επιταχύνουμε λίγο περισσότερο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτό το σημείο. Διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, ειδικότερα αυτή τη στιγμή όπου πρέπει να εγκρίνουμε το συνδέοντα στην Ευρώπη και να δούμε τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά, κατά πόσο αυτά τα χρήματα ενδεχομένω θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια χρηματοδότηση που θα οδηγεί σε πολλαπλουσιασμό των λίγων χρημάτων που έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ερτοκ. Ευχαριστώ κύριε Έχω ένα ερώτημα ε, όσον αφορά την εμπειρία σας από την, πλατφόρμα Λιόν Τωρίνο. Όπως ξέρετε από την νομοθεσία στη Γαλλία, το μέσον ε, των, της πλατφόρμας ε, των διαδρόμων ε, μας περιορίζει όσον αφορά την πρόταση, τις προτάσεις που έχουμε να υποβάλουμε για να προχωρήσει το έργο αυτό με τη βοήθεια του συντονιστή. Εσείς έχετε σε αυτή την πλατφόρμα Λιόν Τωρίνο ε, πολλές πληροφορίες και αξιόλογες εμπειρίες. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε τι εμπειρίες έχετε συλλέξει, τις οποίες μπορούμε στο μέλλον, ελπίζω, να ενσωματώσουμε στο δικό μας νομοθετικό πλαίσιο. Ο Πρόεδρος, πριν από την κυρία Μάισερ, καλώς ορίζω τον κύριο Ρικάρντο από, ε, από το Φριούλι Βενέτσια, από την, Mrs. Ε, Meissner, two minutes. την επαρχία Φριούλι Βενέτσια της Ιταλίας. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ κύριε Μπρίνκος, πολλά ελέγχθησαν για την Ιταλική διασύνδεση από τον κύριο Κάντσια. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι κοστίζει όλο αυτό το έργο με το διασυνοριακό στοιχείο, δεδομένου ότι οι ταλικοσλοβενικές ε, σχέσεις ήταν λίγο δύσκολες. Όλα τα επιστώσεις θα προέρχονται από το ΣΕΦΑ και είναι αφικτή αυτή η χρηματοδότηση. Παραδείγματο χάρη, αν η Ιταλία δεν μπορεί να συμβάλλει τίποτα ή μηδέν, έχει μηδενική συμμετοχή, τι θα γίνει με το έργο. Ευχαριστώ η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ για την ε, έκθεσή σας. Όσον αφορά όλη αυτή την ε, διαδρομή, από ότι αρχίζω εξανατολών. Στη Βουδαπέστη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν χρήματα για το, για το τμήμα που Βουδαπέστη τα σύνορα. Όσον αφορά τώρα τις συνοριακές περιοχές Σλοβενίας Ιταλίας, αυτή η κατάσταση μοιάζει με την κατάσταση Σλοβακίας Αυστρίας. Από ιστορικής ε, απόψεως υπάρχουν και ιστορικά δεδομένα, ένα ιστορικό παρελθόν κλπ. Δυσκολίες. Υπάρχει αυτή η πλατφόρμα των βορειοϊταλικών λιμανιών που επισημούν κάτι άλλο σε αυτή την διαδρομή. Αυτές οι επιθυμίες αλλάζουν τίποτα διότι δεν θέλουν το κόπα. Θέλουν περισσότερο η διασύνδεση να αποβεί προς όφελος των Ιταλικών λιμένων. Δεύτερο, μεταξύ Μπρέσια και Βιτσέντζα. Ξέρω αυτή τη διαδρομή πάρα πολύ καλά και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ολοκλήρωση. Αυτή, δηλαδή η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι πολύ τραβηγμένη στο μέλλον. Και είναι μια, μια διαδρομή που χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τον κόσμο. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες όπως η, το, η πλατφόρμα Λιόν Τωρίνο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εάν αξίζει να επεκταθούμε προς μας ή εάν πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας περισσότερο στα σημεία βάρου στις διαδρομές δηλαδή αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ φορτωμένες. Ο κύριος Βεράνο στην περιφέρεια αυτή συνομιλεί μόνο με τους δικούς του, με τους φίλους του και όχι με αυτούς από τους οποίους πρέπει να επιτύχει συνένεση. Δεν πιστεύω ότι ε, μπορεί να μας βοηθήσει ο συνομιλητής μεταξύ των δύο διαφορετικών μετόπων. Ο άνθρωπος κοιτάει το συμφέρον του και υποστηρίζει τους δικούς του. Η κυρία ε, Βίλς, δύο λεπτά. Εγώ είμαι από το Αμβούργο και έχω μεγάλη εμπειρία από τις μεταφορές βορανότου και βεβαίως αυτός είναι και ο βασικός εμπορευματικός άξονας προς την Νότιο Ευρώπη. Άκουσα ότι σε αυτή τη διαδρομή Λιόν Τωρίνο, δηλαδή από Ανατολή προς Δύση, Ähm, ε, πιστεύω ότι ε, δεν ε, αξίζουν αυτές οι επενδύσεις, δεδομένου ότι οι δαπάνες είναι πάρα πολύ υψηλές. Λιόν, Τωρίνο. Τα, τα κεφάλαια, τα δημόσια κεφάλαια είναι πολύ λίγα και το ερώτημα αν θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την πλατφόρμα δεδομένου ότι δεν προβλέπεται υψηλότερες εμπορευματικές μεταφορές και αντίστροφα από δυσμάς προς Ανατολάς μας θέτει το ερώτημα, αξίζει, αξίζουν τα κονδύλια αυτά. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση ως προς αυτή τη διαδρομή ε, και από τη γαλλική και από την ιταλική πλευρά υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και έχουμε στοιχεία αξιόπιστα από εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση, αλλά με, εκπλήσει, εκπλήττει η αισιοδοξία σας. Μεταξύ Μπολόνιας και Βερόνας η Ιταλία χρειάστηκε 80 χρόνια για τη δεύτερη γραμμή. Και τώρα θέλουμε, να, θέλετε να, να χρηματοδοτηθούν Σλοβενία, Ιταλία, ε, Σλοβα... και, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την παλιά διαδρομή στο Ρίνο. Ε, εντάξει, ας γίνει ένα καινούριο τούνελ, αλλά το κόστος είναι ένα κλάσμα του νέου έργου. Ε, αντί να φτιάξουμε τα κακώς κείμενα και να τα βελτιώσουμε, θέλουμε να κάνουμε, ξεκινήσουμε καινούρια λίγα δαπανηρά έργα. Τι, τι θα κάνετε όταν συναντηθούν στις 3 Δεκεμβρίου ο Μόντι με τον Ολόν και ο Ολόν πει δεν έχω λεφτά φράγκο δηλαδή. Και ο Μόντι πει ότι, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι οι τράπεζες εποφελούνται από όλα αυτά τα έργα και βάζουν λεφτά στην τσέπη τους και ο Μόντι πει όχι αυτό θα γίνει. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα χρειαστώ καν δύο λεπτά. Uh, between and Slovenia. Θέλω να ρωτήσω για τον άξονα Ιταλία-Σλοβενίας που δεν θα είναι μόνο για εμπορεύματα αλλά και για επιβάτες. Τι θα γίνει όταν θα προσπαθήσουν να έχουν διασυνοριακή σύνδεση συντεριές, τι δεν υπάρχει τίποτα, καταφτάνουν τουρίστες ε, να επισκεφθούν ε, είτε τη Σλοβενία, είτε τη Βόρεια Ιταλία, είτε και την Κροατία και στην ε, περιοχή φτάνουν στη, από τη Βενετία, από τη Βερόνα, στα αεροδρόμια της Τεριέστης και μετά προσπαθεί να πάει κάποιος στη Σλοβενία, φτάνει στην Τεριέστη, έχει τρία λεωφορεία την ημέρα θα υπάρξει κάποια διασύνδεση ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εξίσου και για εμπορεύματα και για επιβάτες αυτή η διαδρομή και πού θα μπορεί κάποιος να κάνει απόβαση επιβίβαση. Θα μπορεί να πάει απευθείας από το Μιλάνο στη Λιουμπλιάνα χωρίς να σταματήσει. σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί τοπικό πρόβλημα στην Τεργέσπη, ιδίω ε, από τουρίστε που απλώς περνούν από την περιοχή. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση και από μένα, κύριε Μπρίνκχορστ. Ένα από τα πράγματα τα οποία με χαροποιεί ε, να βλέπω ε, είναι ότι υπάρχει και η σύνδεση με το κόπερ, γιατί το κόπερ είναι το μόνο μέρος στο οποίο πραγματικά ε, τα όσα εκφορτώνονται στο λιμάνι μεταφέρονται μέσω αυτοκινητοδρόμων και χαίρομαι που περιλαμβάνεται γι' αυτό. Θα θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα είναι ευχαριστώ να απαντάει κανείς σε πολλές ερωτήσεις, ε, ειδικότερα ερωτήσεις που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ας ξεκινήσω με τη γενική ερώτηση του κυρίου Κράμαρ, διότι σας έχω και ακριβώς μπροστά μου. Μετά από πολλά χρόνια στην πολιτική έμαθα να μην απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις. Θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα όταν χρειαστεί. Εάν στις 3 Δεκεμβρίου δεν υπάρχει συμφωνία θα έχουμε μια νέα κατάσταση. Εγώ όμω είμαι αισιόδοξο που είμαι Ευρωπαίος και εσείς είστε Ευρωπαίος και θα χρειαστεί να είστε αισιόδοξο. Και πιστεύω πραγματικά ότι ο κ. Ολάντ και ο κ. Μόντι δεν είναι ανόητοι. Και αυτό απαντά και την ερώτηση της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Εάν δύο χώρες που εμπλέκονται άμεσα μετά από πολλούς προβληματισμούς, με πολλές δυσκολίες χρηματοδοτικές, είναι έτοιμες να επικυρώσουν με νέα συνθήκη και να επιβεβαιώσουν ότι για στρατηγικούς και άλλους λόγους ο τουρισμός είναι σημαντικός, ποιος είστε εσείς και ποιος είμαι εγώ να τις κρίνουμε αρνητικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι. Μετά από τις συζητήσει που είχαμε, ε, κύριε Λίχτεμπεργκερ, και πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εν τέλει εκεί. Και μετά θα την επικυρώσουμε φυσικά και μετά θα έχουμε ένα νέο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις του τι θα συμβεί εάν καθίστανται απερχαιωμένες στις 4 Δεκεμβρίου και ευχαριστώ θα έρθω αν θέλετε σε μια δική συνάντηση ε, μαζί σα στις 4 Δεκεμβρίου για να σα πω τι θα γίνει μετά από την επικύρωση αυτή τη απόφαση. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω πρώτα στον κύριο Καντζάνο, όπω Καντζιάνο. Κατσιάν. Πάντα είναι ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει σα. Ε, έχουμε και εκείνη την ιστορική γραμμή που αναφέρατε. Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα μπρόσβο να χρησιμοποιήσουμε τις συνδυασμένε μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα επανέλθω σε λίγο στα, στα ε, λιμανιά της Βορειάς Αδριατικής διότι δεν υπάρχει αντίθεση εκεί και φυσικά θέλουμε να προωθήσουμε τις συνδυασμένε μεταφορές και εκεί. Αλλά όπω είπα για ιστορικούς λόγου, ίσω χρειαστεί λίγο περισσότερο καιρό. Ένα κομμάτι της γραμμή είναι. Έχει μπλοκαριστεί Είχα μια συζήτηση σήμερα το πρωί με έναν από του υπουργού τη περιφέρεια, του ονομάζουμε υπουργού, γιατί οι περιφέρειε που γνωρίζετε στην Ιταλία είναι πολύ σημαντικέ και μιλήσαμε για ένα κομμάτι τη γραμμή που δεν είχε σχέση με την περιοχή που διέρχεται από τα σύνορα, αλλά ένα κομμάτι τη Ιταλία στο Νότο. Και με ρώτησαν κατά πόσο θα ήταν ωφέλιμο για μένα να συνεργαστώ και να βοηθήσω, διότι υπάρχουν δυσκολίε στο εθνικό πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι πριν κρίνουμε και πούμε ότι ένα κράτο πάντα τα κάνει όλα καλύτερα. Πολλέ φορέ προτιμούν μια ευρωπαϊκή συνεργασία. Γι' αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά αν δεν υπάρχουν χρήματα για εθνικά προγράμματα, μπορούμε να βοηθήσουμε με εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία. Το ζήτημα των ομολόγων για προγράμματα, έργο, εκτέλεση έργων, ε, των project bonds, είναι δημόσια χρήματα φυσικά. Πιστεύω για τη Σλοβενία και την Ουγγαρία θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να επανεξετάσουμε το ζήτημα. Τώρα, η εμπειρία μου είναι πολύ θετική. Για ποιο λόγο, διότι επιτρέπει στην Κομισιόν και σε μένα ως συντονιστή να κινηθώ πέραν των κυβερνητικών δομών γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι της Λιών, διότι έχουμε το Transalpine στη Γαλλία που συνδυάζει όλες τις μεγάλες εταιρείες επιμελητίας υποδομών και παραγωγής που ενδιαφέρονται για αυτή τη γραμμή και στην Ιταλία υπάρχει το Transpandana. Αυτοί μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και το ίδιο ισχύει και για τις ίδιες περιφέρειες και μάλιστα ο κύριος Μίλανο έχει πάντα παίξει επικοδομητικό ρόλο σε αυτές τις συναντήσεις κατά την απόψή μου. Λοιπόν η ιστορική γραμμή δεν θα μπορούσε να έχει αποκατασταθεί τόσο γρήγορα εάν δεν είχε εξασκηθεί πίεση από την πλατφόρμα και τους συμμετέχοντες της. Κύριε Μάισνερ. Μάισνερ, στην περίπτωση του Κόπερ τα χρήματα δεν είναι το σημαντικότερο. Διότι για τους Σλοβαίνους είναι πολύ σημαντικό να έχουν απευθεία σύνδεση μεταξύ του ενός λιμανιού που έχουν στην Αδριατική και και της ενδοχώρα. Δεν είναι ρεαλιστικό να, χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιείται αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Καθώς θα αναπτύσσεται η τριγέστη και το κόπερ, δεν θα υπάρξει κανένας τρόπος διαφυγής. Θα υπάρξει περισσότερη εναρμόνιση στην Αδριατική. Πριν πολλά χρόνια, όταν εργαζόμουν στις κατοχώρες, ε, από προέρχομαι, συζητήθηκαν ε, πολύ το Ρότερνταμ και η Τεργέστη. Υπήρχε σύνδεση, υπήρχαν μεταφορές από τους σιδηροδρόμους στα πλοία, οι οποίες σταμάτησαν λόγω αναποτελεσματικότητας μέσα στον χρόνο. Πιστεύω έντονα ότι αν η Βενετία, η Τεργέστη και το Κόπερ συνεργαστούν και τα λιμάνια της Βόρειας Αδριατικής αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τη Γένοβα, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για την αυξανόμενη κυκλοφορία προς την Ανατολή, προς την Κίνα και άλλα μέρη, διότι πιστεύω αυτό είναι το μέλλον. Και αυτό είχα πει και στην εκστρατεία για το κόπερ. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, απάντησα ήδη στα θέματα Λιοντουράν, αλλά για τη Βουδαπέστη. Ναι, φυσικά δεν υπάρχουν χρήματα στη Βουδαπέστη. Αλλά όπως γνωρίζετε, τον κύριο Χέρσταν, θα περάσω στα γερμανικά κύριε Πρόεδρε. Ήταν πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν και είπε ότι υπάρχουν πραγματικότητες τις οποίες μπορούμε να παραμερίσουμε. Δηλαδή υπάρχουν ε, ιστορικά, ιστορικές πραγματικότητες που μπορούν να παραμεριστούν. Εάν δεν είχε εκείνος αρχίσει, δεν θα ήμασταν στη θέση που είμαστε σήμερα. Κάποια φορά λοιπόν χρειάζεται η αισιοδοξία. Δεν χρειάζεται απεσιοδοξία. Και υπάρχει και υπάρχουν ιστορικές πραγματικότητες που μπορούν να αλλάξουν στη Βουδαπέστη. Είναι σαφές ένα πράγμα. Η Βουδαπέστη ιστορικά ήταν η καρδιά του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως η Βιέννη. Και θέλουμε να το αυξήσουμε αυτό. Το θέμα της έλλειψης πιστώσεων δεν σημαίνει ότι τα πάντα θα νεκρωθούν και δεν θα λειτουργήσουν πρέπει Βουδαπέστη, Σλοβενία να αρχίσουν να συνεργάζονται. Ε, δεν είναι φρούδα η υπόσχεση αυτή, είναι η πρόθεσή μας. Διαφορετικά, ας αλλάξετε συντονιστή. Επίσης, το, ο κόμβος της ε, Βόρειου Ιταλίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και συζητώ και με άλλους συντονιστές για τα οδικά δίκτυα. Είναι πολύ σωστό να έχουμε μία συνάντηση μεταξύ του Κόπερ, της ε, Τεργέστης και της Βιέννης για να δούμε τι θα γίνει με τη γραμμή προς ε, Βορρά. Όσον αφορά τώρα το τμήμα Μπρέσια Βιτσέντζα, Ξέρω τις δυσκολίες, ως συντονιστής δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα, αλλά θα περάσω τα προβλήματα αυτά και τις θέσεις σας ε, στους ε, διαχειριστές αυτής της, ε, του τμήματος. Και το, η άποψη του κυρίου Βεράνου και η δικιά μου διαφέρουν. Εκείνος είναι συντονιστής <laughs> της Ιταλικής πλευράς και είχε 180 συναντήσεις. Ε, δεν μπορείτε να πείτε λοιπόν ότι και οι 180 συναντήσεις ήταν μόνο με δικούς του φίλους και ανθρώπους. Ε, η, κυρία Βίλς, ναι. Ε, σας παραπέμπω στο ίδιο ερώτημα. Οι κύριοι Μόντι και Λάοντ θα συναντηθούν στις 3.12 εάν δεν συμφωνήσουν ή η, συμφωνία την κρίνεται απέσια, αυτό αφορά εκείνους και όχι εμένα. Και τέλος, το θέμα Ιταλίας-Σλοβενίας. Ρωτάτε πού θα αποβιβάζεστε. Θέλετε να πάρουμε ένα τρένο μαζί. Όταν πηγαίνετε στην Τεργέστη με τρένο, μπορείτε να κατέβετε στην Τιβάτσα, στη Λουμπλιάνα ή στο Μάριμπορ ή στο Μπούμπα ή στη Βουδαπέστη. Αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Οκτώ ώρε και δεν ξέρω αν θα αντέξετε να κάθεστε μαζί μου. 8 ώρε στο τρένο. Κύριε Πρόεδρε, αυτές ήταν οι απαντήσει που είχα να δώσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ας μην μπούμε σε περιγραφή των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπρινκχόρς. Θα ακολουθεί ο κύριος Πατ Κόξ με το έργο προτεραιότητας αριθμός 1 και έχετε και το επίμαχο ζητήματα του Brenner Base ε, της σύραγγας αυτής. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Όπω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σα υπέβαλα μία γραπτή έκθεση 23 σελίδων. Δεν θα τη διαδρέξω όλη βέβαια τώρα. Θα ήθελα επίση να ζητήσω τη γραμματεία σα κύριε Πρόεδρε να διανύμει ένα σύντομο DVD, το οποίο είναι διαθέσιμο για λόγους ενημέρωσης προς τα μέλη, αλλά ε, επίσης ε, διαβιβάζουμε και τα όσα συνέβησαν ε, με τη σύραγγα, οπότε είναι ε, ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που σας δίνει πληροφορίες. Ήταν πρόκληση η φετινή χρονιά και θεωρώ όμως ότι συνοπτικά κάναμε συνεχή πρόοδο. Και η Αυστρία και η Ιταλία έχουν προγράμματα λιτότητας. Παρόλα αυτά όμως και οι δύο χώρες, κάτι για το οποίο είναι αξιέπαινες, δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν με πολύ σημαντικά ποσά επιπλέον χρηματοδότησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Για την Αυστρία υπάρχει εγγύηση για πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από σήμερα μέχρι το 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος και για την Ιταλία έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ ε, μέχρι το 2015 με επιπλέον 300 εκατομμύρια που εκκρεμούν ε, για την περίοδο αυτή. Και οι δύο κυβερνήσεις, και η Αυστριακή και η Ιταλική, ε, όσον αφορά τη σύραγγα Μπρένερ ε, Μπρέσε και τους ε, ε δρόμους της νότιας πρόσβασης έχουν αποφασίσει να επανασυστήσουν την Διακυβερνητική Επιτροπή που αρχικώς θα έπρεπε να ξεκινήσει για, την, για τη σύραγγα του Brenner Base αλλά από εκεί και πέρα ε, θεώρησαν ότι υπάρχει χρησιμότητα για να συνεχιστεί αυτή η διακυβερνητική και διαπεριφερειακή ε, σχέση που υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης για τη μελλοντική χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και βάση του κείμενου προϋπολογισμού και να προγραμματίσουν και μελλοντικά κονδύλια. Τι έχει γίνει μέχρι τούδε. Όσον αφορά το η σύραγγα Brenner Base έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα 24 χιλιόμετρα ε, σύραγγας μεταξύ ε, παράπλευρες πρόσβασης ε, ε, τούνελ που υπάρχουν για να μπορέσουμε να έχουμε σύνδεση και στις δύο πλευρές, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ένα διερευνητικό τμήμα σύραγγας και επίσης ένα τμήμα ε, της έχει ξεκινήσει, 45 ε, μέτρα έχουν γίνει μόνο, αλλά είναι το πιο ε, σημαντικό από πλευράς γεωλογίας ε, και η πρόοδος γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετική θα μπορέσουμε να έχουμε επιπλέον 2,4 χιλιόμετρα σύραγγας στη συγκεκριμένη περιοχή ε, σε μία από τις, με μία από τις παρούσες συμβάσεις και το τελευταίο τμήμα της σύμβασης για το τελευταίο κομμάτι της σύραγγας ε, θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Συνοπτικά λοιπόν, ναι μεν υπάρχει λιτότητα, αλλά υπάρχει συνεχής ε, και ενεργός δέσμευση μεταξύ των κρατών μελών και των βασικών ενδιαφερομένων για το συγκεκριμένο πρόσβαση. Τώρα, για τη διαδρομή βόρειας πρόσβασης Αυστρίας-Γερμανίας από το Ίνσπρουκ ε, στο Μόναχο. Εκεί έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος. Εχθές είχα το προνόμιο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραστώ στα εγγένεια της ε, κάτω γραμμής, ένα τμήμα 40 χιλιόμετρων μεταξύ ε, Αυστρία στη βόρεια πρόσβαση και υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε αυτό το σημείο. Υπάρχει επιπλέον ασφάλεια και συμβατότητα. Ε, είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη γραμμή της κοιλάδας του κάτω τμήματος. Ο υπήρχαν οι αρμόδιοι υπουργοί από την Αυστρία και τη Γερμανία οι οποίοι υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης και κατόπιν ε, μετά την υπογραφή του μνημονίου τον Οκτώβριο ε, το Υπουργείο στο Βερολίνο υπέγραψε για χρηματοδότηση για τα δίκτυα των σιδηροδρόμων τη Γερμανία, για να ξεκινήσουν συνεργασία με την Αυστρία για να ξεκινήσει ο σχεδιασμό του επόμενου σταδίου. Και ελπίζουμε ότι αυτέ οι εργασίε θα βοηθήσουν και θα υπάρξει περαιτέρω πρόεδρο στι επόμενε εβδομάδε και θα υπάρξει και πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη μελλοντική ε, ανάπτυξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Για την νότια πρόσβαση τώρα μεταξύ ε, Ιταλίας και Βόρειας ε, και Νότιας ε, ε, Αυστρίας, ξέρετε ότι αυτά είχαν καθυστερήσει, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η πρόοδος, έχει ξεκινήσει το πιο περίπλοκο ζήτημα μεταξύ Φορτέτσα και Πόρτε Γκαρντένα, από την ε, Επιτροπή Δημοσίων Δαπανών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα λοιπόν έχουν δοθεί ένας προκαταρκτικός ε, προϋπολογισμός 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Περιμένουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες όσο προχωρούμε και είμαι αισιόδοξο ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει λιτότητα, η δέσμευση των αρχών να υλοποιήσουν τα έργα αυτά υπάρχει. Όσον αφορά τώρα ένα κονδύλιο 550 εκατομμυρίων ευρώ ε, διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δημιουργείται υπό την αιγίδα του οργανισμού που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο Α28 στην Ιταλία για την περιοχή του Τρέντο ε, που έχουν ενδιαφέρον για τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα διατεθούν για το πρόγραμμα, αλλά προσπαθούμε να ε, δούμε πώς θα διεξαχθεί αυτή η πολύ ιταλική συζήτηση για το πώς ε, θα διασκεδάσουμε τις παραδοσιακές ανησυχίες για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Όσον αφορά το τμήμα Βερολίνο-Μόναχο, λογικά θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2016 και εντός της Ιταλίας ε, όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί το κατώτερο τμήμα ε, της κοιλάδας ε, Αυστρίας-Ιταλίας, ε, επομένως τα βασικά τμήματα έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης θα έχουμε και χρηματοδότηση από το Συνδέοντα στην Ευρώπη, το Connecting Europe και ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσατες δεν υπάρχει ανάγκη να σχολιάζουμε πριν ολοποιηθούν κάποια πράγματα. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα πολιτικής εδώ για το πώς θα κατανεμωθούν τα κονδύλια και εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεγιστοποιήσουμε και τα διασυνοριακά τμήματα. Και γιατί σας το λέω αυτό. Διότι αν εξετάσετε όλους τους χάρτες ε, όλων των ετών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών ε, ε, δικτύων, τα σημεία που λείπουν, οι σύνδεσμοι που λείπουν είναι τα διασυνοριακά τμήματα και αν θέλουμε να συνεισφέρουμε κάτι, αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Όσον αφορά τώρα, κύριε Πρόεδρε, του υπόλοιπου τομεί πολιτική, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να υπάρξει περισσότερη πρόοδο και να μπορέσουμε να οργανώσουμε ε, λίγο καλύτερα τις μεθόδους εργασίας μας για μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εάν ε, δημιουργήσουμε κατάλληλες ιδιοδρομικές υποδομές και ε, με χαρά θα ήθελα να σας πω εδώ ότι μετά από την πρωτοβουλία που είχαμε να συνεργαστούμε με τον γερουσιαστή Ντίνη και τον πρόεδρο του ε, ε, της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον κύριο Φίνη. Η Ιταλία έχει πλέον κυρώσει τη σύμβαση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κανονικά το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα για να πιέσετε το θέμα αυτό περαιτέρω. Γιατί γίνεται αυτό, Γιατί όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη έχουν συμφωνήσει να τηρηθούν κάποιε αρχέ που θα μα δώσουν ένα πλαίσιο προκειμένου να αναπτύξουμε ε, και να προσδώσουμε ουσία στα συνοδευτικά μέτρα. Αλλά υπάρχει και μία περιοχή ε, γύρω από τις Άλπεις και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε επίπεδο περιφερειών και πώς αναπτύσσονται τα σημεία αυτά και θα πρέπει να συνδέσουμε ε, τις ε, ενδοκρατικές ανησυχίες που υπάρχουν για τις ε, Άλπεις με τις ενδοπεριφερειακές ανησυχίες που υπάρχουν για τις περιφέρειες, να γίνει κατάλληλη παρακολούθηση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όσον αφορά τώρα την πλατφόρμα για τον διάδρομο του Μπρένερ, αυτή η δράση συνεχίζεται και ε, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τις προτάσεις μας για τα συνοδευτικά μέτρα. Η πρότασή μου, η αίσθησή μου είναι ότι γίνονται πάρα πολύ καλά ε, πράγματα από πλευράς ε, γεωλογικών, υδρολογικών και χρηματοδοτικών θεμάτων, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο στο λογιστικό, όπως το αποκαλώ αυτές τις δέσμεις ε, διαδρόμων. Έχουμε πέντε περιφέρειες, ε, πάρα πολλές ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ο καθένας έχει διαφορετικές ε, προτεραιότητες στα συνοδευτικά μέτρα και στο θεματολόγιο τους. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπτύσσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο για να προχωρήσουν με λίγο πιο τυποποιημένο τρόπο. Και αυτό θα προχωρήσει όχι μόνο με τα όσα κάνουμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα για τις επενδύσεις, αλλά και με τον κανονισμό για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει η δυνατότητα βάσει των ε, κείμενων κανόνων να έχουμε μια νέα σύραγγα που θα εξοικονομεί χρόνο μισή ώρα μόνο από αυτή τη σύραγγα και επειδή δεν θα υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση, κάποιο ο οποίο θα κατεβαίνει από το τρένο, θα περπατάει 700 με 700 μέτρα μέχρι ε, ε, την άκρη, θα χάνει το φανάρι και θα χάθουν όλες οι εργασίες που κάνουμε για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Και τι γίνεται αυτό από μία νοησία. Και κάποιος πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να αρχίσει να εργάζεται αυτή τη στιγμή, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα όσα γίνονται ε, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση, αντλώντας διδάγματα από το Στοντγκάρ 21 και τα όσα συνέβησαν εν γέννη. Ε, και στο, συναντήθηκα με τους δημάρχους στο Νότιο Τυρόλο, με το Τρεντίνο, μίλησα και με κάποιους υπευθύνους των προγραμμάτων ε, στην περιοχή και προσπαθούμε πραγματικά να είναι όλοι μαζί μας. Γιατί ένα από τα βασικά διδάγματα που μαθαίνουμε είναι ότι για τις επενδύσεις, για τις υποδομές είναι ότι οι πολιτικές εναλλακτικές λύσεις ε, στην αρχή ενός προγράμματος, ακόμα και αν είναι θετικές, μας κοστίζουν περαιτέρω χρόνο. Και επομένω, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, η αρχική πατρότητα, η μητρότητα του προγράμματο μπορεί και να χαθεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να χαθούν τεράστια προγράμματα επειδή υπάρχει πρόβλημα πολιτική επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη πολιτική επικοινωνία και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να έχουμε ως στόχο να έχουμε αποτελέσματα. Υπάρχουν ε, κάποιες ερωτήσεις που ακούστηκαν προηγουμένως για να σας προλάβω για τα ομάλογα έργου στο μέλλον και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Εχθές στην Αυστρία όταν ξεκίνησε η συζήτηση ε, η Επιτροπή υπέγραψε μια συγκεκριμένη ε, δραστηριότητα για την ε, ε, χρηματοδότηση και το EIP έχει ήδη κάνει επέκταση μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Για το πρόγραμμα του Brenner λοιπόν θα προτιμούσαμε να είχαμε κάτι το οποίο θα έχουμε μετά από το CEF για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ομόλογα έργου ή κάτι αντίστοιχο. Για να αναπτύξουμε λοιπόν κατάλληλες μεθοδολογίες, να έχουμε κατάλληλη οργάνωση και να έχουμε δυνατότητες επικοινωνίας για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτά τα προγράμματα και να έχουμε και τις κατάλληλες δυνατότητες στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τέλος, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είπα και πέρσι, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ καλή βοήθεια από τον κύριο Λέο Χούμπερτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς τη βοήθειά μου, το, τη του έργο μου θα ήταν άχρηστο. Ευχαριστώ κύριε Κόξ και καλώς ήρθατε στο, στον κόσμο το, της δυστυχίας των τρένων που είναι ο δικός μου. Ο κύριος Κάντσαν, δύο λεπτά παρακαλώ. Και όχι, τα, τα ομόλογα έργα έχουν απαντηθεί. Δύο λεπτά ο κύριος Κάντσαν. Εκτός μικροφώνου ο μιλήτης. Ευχαριστώ κύριε Πατκόξ για το έργο σας εξαιρετικά δύσκολο. Το κατανοώ ωστόσο. Μία ερώτηση που έκανα πριν δεν απαντήσατε. Η ερώτησή μου ήταν η αργοπορία οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων, στα προβλήματα επιτόπου, επειδή δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για το τι θα κάνουμε. Είναι κάτι δηλαδή ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οφείλεται στην ελάχιστη εξουσία που έχετε εσεί για να διαχειριστείτε αυτό το έργο. Η δεύτερη μου σκέψη είναι ότι εγώ λέω αν είχαμε διαθέσιμα τα χρήματα σήμερα εδώ για να μπορούμε να υλοποιήσουμε έργα κατά την άποψή σας είναι βιώσιμο το έργο αυτό από οικονομική, περιβαλλοντική και εδαφική άποψη επιτόπου και από κοινωνική άποψη. Διότι από όσο κατάλαβα μιλάμε πολύ για τις οικονομικές δυνατότητες που φυσικά αποτελούν ένα πρόβλημα αλλά τείνουμε να ξεχνάμε τα προβλήματα βιωσιμότητας και εδαφικής συμφωνίας. Αυτή είναι η δική σας λειτουργία Είστε ικανοποιημένοι με τις εξουσίες που έχετε, είναι επαρκείς ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση, διότι την επόμενη εβδομάδα θα πάμε να κάνουμε μια άλλη δουλειά και τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Κυρία Μπιλμπάου, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Κόξ. και μας ανέφερε την εξέλιξη του έργου, επεσήμανε δύο πράγματα που κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα απ' όλα τα προβλήματα που οφείλονται στο ε, διάφορα στάδια ενός έργου και στο γεγονός ότι αφορά πολλές διαφορετικές περιφέρειες η ανάγκη συνέχιση με αυτή τη γραμμή, καθώ και το να λάβουμε υπόψη ότι θα χρειαστεί να ορίσουμε προτεραιότητε, ε, να δώσουμε προτεραιότητα σε προγράμματα προσθέμενες αξία με περιορισμένο προπολογισμό. Τώρα, εσεί είπατε, παρακολουθείτε το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη, τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και υποθέτω λοιπόν ότι ακολουθείτε και τι κατευθυντήριε γραμμέ. Τώρα, έχοντα ακούσει όλου του συντονιστέ, ε, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο να αυξήσουμε τον αριθμό έργων προτεραιότητας όπως ορίζονται στι κατευθυντήριες γραμμέ. Και και τι θα συνέβαινε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσιζε να εγκαταλείψει τη Μεθολογία συμπεριλήψης έργων. Συμφωνείτε ότι η Ευρώπη έχει διευθετήσει αυτά τα διασυνοριακά θέματα που υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες. Μόλις μιλήσατε για την ανάγκη να ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές, να ορίζουμε εναρμονισμένες μεθόδους εργασίας. Όσον αφορά αυτό, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τι συμβάσει προγραμμάτων που πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ όλων των κρατών μελών σε σχέση με αυτά τα έργα. Κύριε Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Κόξ για την έκθεση σας. Τουλάχιστον είπατε ένα λόγο, μία πρόταση για τα συνοδευτικά μέτρα ε, όταν μιλάμε για τη μετάθεση προς τις συνδρομικές γραμμές, ενώ οι άλλοι συντονιστέ δεν είπαν τίποτα. Ε, δεν γίνεται λοιπόν αυτό από μόνο του, όπως το ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτή η μετατόπιση, αυτή η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο με την ύπαρξη συνοδευτικών μέτρων. Όμως εδώ στο Νότο τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Πρώτον, οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι ε, καταργούν χρονοθυρίδες για τις σιδηρομικές γραμμές ε, στις ε, εμπορευματικές μεταφορές διότι θέλουν να δώσουν το βάρος στις ε, μεταφορές, στις μεταφορές επιβατών. δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν κίνητα ε, για να αυξηθούν οι εμπορευματικές μεταφορές και να μετατοπιστούν, να μεταφερθούν από τους οδικούς άξονες στους σιδηροδρόμους. Έτσι λένε. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα ότι αυτή τη στιγμή οι κατευθυντήριες γραμμές της Ιταλίας βασίζονται στη σύμβαση και αυτά τα δύο στοιχεία της βελτίωσης των μεταφορών και την ε, διεύρυνση της χρήσης της, ε, της Eurovignette είναι πολύ θετικά. η, νότια πρόσβαση, η πρόσβαση στις νότιους άξονες, εκεί δεν συμμερίζουμε την αισιοδοξία σας. Όταν κατεβαίνω από το Στρασβούργο στη Βόρεια Ιταλία, Οι ήδη υπάρχ, τα ήδη υπάρχοντα τμήματα στην Ελβετία δεν προεκτείνονται προς την Ιταλία, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση του δυναμικού. Και τονίζω και πάλι, εμείς εργαζόμαστε για την πολιτική των μεταφορών και όχι μόνο για την πολιτική κατασκευών. Και τέλος, όταν κατασκευάζουμε κάτι το οποίο είναι συνεχή, δεν χρησιμοποιείται, ε, όπως έγινε στην Αυστρία, το πρόβλημα οξύνεται. Ο κύριος ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και η έντονη διαβούλευση είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, το θέμα είναι υπάρχει ανταγωνισμός ε, μεταξύ Γένοβας Ρότερνταμ ε, έχουμε ένα μοντέλο ήδη με το τούνελ του Λότα. Ε, υπάρχει και, και ανατολικό, ανατολικά έχουμε το τούνελ Brenner Base 1 και Brenner Base 2. Ε, υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός στους δύο Ανατολή Δύσεως. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να τύχουμε της χρηματοδοτικής απαλληγής και υπό το πρίσμα της του στις, ε, στο συνεδρίο της ΔΟΧΑ ε, της σύσκεψης της ε, διάσκεψης ΔΟΧΑ για το περιβάλλον, πρέπει να ξέρουμε το, την κατανάλωση ενέργειας αναεπιβάτη Γι' αυτό πρέπει, έχοντα υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία περιβαλλοντικά, ανταγωνισμού κλπ, να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Και πώς θα, διαχειριστείτε το συντονισμό του, του, το 21, οδική άξονες στη θάλασσα, οδική χάρτες θαλάσσης. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ, το έχουμε συζητήσει το θέμα και είπατε ότι εδώ κάνουμε μπαλώματα στους σιδηροδρόμους. κουρελού δηλαδή έχει γίνει το θέμα. Και σας ρωτώ, η, η προτεραιότητά μας είναι ένα μεγάλο έργο με το οποίο μπορούμε να επαναδραστηριοποιήσουμε διάφορες διακλαδώσεις μεταξύ Γερμανίας, Πολωνίας τα τελευταία 23 χρόνια μία νέα γραμμή, ένα νέο τμήμα έχει γίνει. Δεν θα πρέπει να δώσουμε βάρος στο, στην τελική ε, ε, φάση του έργου εκεί, δηλαδή που σταματάει το έργο και όχι μόνο εκεί που ξεκινάει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ε, ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για τις γραμμές στην πρώην Ανατολική Γερμανία, αλλά έχουμε διακόψει την Ιένα, ε, την Λιψία, έχουν κοπεί ε, αυτοί οι σταθμοί. Δεν έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή και επομένει ο πληθυσμός. Και το ήταν. Το δικό σας έργο τελειώνει στο Βερολίνο. Όμως, νοτίως του Βερολίνου υπάρχουν διασυνδέσεις η διασύνδεση Βερολίνου στο Χόλμις διαμέσου του Ρόστοκ Βαρνεμούντε, γιατί δεν τη λαμβάνεται υπόψη αυτή. Μήπως ε, ε, πρέπει να πάει κανείς να κάνει μια παράκαμψη 130 χιλιόμετρα μέσω Αμβούργου για να φτάσει στη Στοχόλμη. Γιατί δεν ακολουθείτε τον άξονα, ε, γιατί κοιτά, δεν κοιτάτε και άλλους διαδρόμους και όχι μόνο το Βερολίνο. Ο κύριος Κόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Κάντσιαν, η ερώτηση για, το, προ, προ, για την πρόοδο επανερχόμαστε στο αν το ποτήρι είναι μισοάδιο μισογεμάτο. Σας είπα ότι είναι μεγάλο πολιτικό επίτευγμα το ότι πείσαμε όλους τους βασικούς παίκτους να επενδύσουν δύο δισεκατομμύρια, όχι λιγότερο από δύο δις, στο, στο μέσο μιας ε, της σημαντικότερης κρίσης λιτότητας που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να απαντήσω. Και για το τα, τα ωφέλη αυτού του έργου δεν έχω εδώ αντίγραφο, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε στον πρόεδρό σας όσον αφορά το τούνελ αυτό του Μπρένερ, υπάρχουν μέσο πρόθεσμα και βράχη πρόθεσμα ε, πολλά πλεονεκτήματα στη φάση αυτή κατασκευής. Έχουν σημειωθεί, έχουν επισημανθεί τα πλεονεκτήματα ακόμα και στη φάση αυτή την βραχυπρόθεσμη και μέσο πρόθεσμη της κατασκευής. Όλοι θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την, ε, τα, τις επιπτώσεις αυτών των έργων. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Άλπων θέλουμε να μειώσουμε την, ε, τις, εκπομπές, τη ρήπανση, τους θορύβους κλπ. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αναπτύξουμε τα συνοδευτικά μέτρα με την ίδια ένταση με την οποία αναπτύσσουμε την υποδομή. Διαφορετικά επενδύουμε κατά μη ικανοποιητικό τρόπο, κατά ελάχιστα ικανοποιητικό τρόπο. Και πιστεύω ότι αυτά τα συνοδευτικά μέτρα από που βγουν πιο ωφέλιμα από την καθ' αυτό κατασκευή της, ε, ανάπτυξη της υποδομής. οι, πολλές φορές η υποδομή ενσωματώνει ε, υψηλή τεχνολογία και σε έναν πανέμορφο μέρος της Αυστρίας σε 41 χιλιόμετρα, λίγο πανερό, αλλά το επίπεδο της ενσωμάτωσης του έργου αυτού με την τοπική ε, ε, με το τοπικό περιβάλλον είναι εξαιρετικό. Είναι η, η είναι σε μια κοιλάδα το έργο αυτό και όσον αφορά το, τις κατευθυντικές γραμμές του CEF παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τι συζητήσεις στο Συμβούλιο και ο ρόλος μου είναι να παρακολουθώ όλες αυτές. Α, για το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά εγώ περισσότερο κοιτάω τις ε, συγκεντρώσεις των ελληπαντών και δεδομένου ότι έχετε έρχονται και τα Χριστούγεννα, πρέπει να δούμε τι θέλουμε μεταξύ αυτό που είναι διαθέσιμο και μεταξύ της ιδανικής Ευρώπης. Ε, πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα μαζί με το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να ε, βρουν τη σωστή ισορροπία. Όσον αφορά στο, τα, τις συμβάσεις, το BBTSC, έχουμε ε, εταιρείες ε, αυστροϊταλικές ε, υποδομών, εταιρείες υποδομών που εκπροσωπούν την πρώτη γραμμή των επενδύσεων των χωρών τους και αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται πάρα πολύ καλά μαζί τους. Για το μοντέλο του Brenner, είναι, το μοντέλο του Brenner είναι πρωτοπόρο για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία για να διαμορφώσει ένα αποδεκτό πλαίσιο και στις, στα δύο συμβαλόμενα μέρη. Επίσης, σε αυτά που είπε η κυρία Λίχτενσταν, συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, 11 cents ανά χιλιόμετρο είναι το κόστος, στην Αυστρία 68 cents ανά χιλιόμετρο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και υπάρχει μεγάλη απόκληση στις προτιμήσεις του κόσμου. Δεν ξέρω ε, αν αυτά τα συνοδευτικά μέτρα είναι καλά ή άσχημα όσον αφορά το υψηλό ή το χαμηλό κόστος. Αλλά στην Αυστρία το κόστος αναλύτρου ντίζελ είναι χαμηλότερο διότι υπάρχουν λιγότεροι ειδικοί φόροι. Οπότε, οι περισσότεροι θα, προτιμήσουν ορθολογικά το τούνελ του Μπρέμερ του διότι το κόστος είναι χαμηλότερο και ε, θα είμαστε ανέντιμοι εάν ακολουθούμε μόνο τις, ε, την τιμολόγηση ως κατευθυντή γραμμή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το κόστος είναι χαμηλότερο του Μπρέμνερ. Σχετικά με την χρηματοδότηση των Ελβετών στη σκανδιναβική διασύνδεση, ε, εγώ προσπαθώ να σε εξηγήσω εμείς τι κάνουμε για να προωθήσουμε αυτές τις επενδύσεις. Πρώτον, οι επενδύσεις μας θα πρέπει να, έχουν, να είναι λογικές, ορθολογικές και πρακτικές. Δεύτερον, πρέπει να αποκρίνουν τις περιβαλλοντικές ανάγκες και να είναι ε, βιώσιμες και αηφόρες με την πάροδο του χρόνου. μπορούμε, όπως ρώτησε ο κύριος Κάμερ, αντί να ακολουθούμε μία, ένα μεγάλο έργο, να αναπτύξουμε περισσότερα μικρά έργα και δίκτυα. Μήπως αυτή είναι μία καλύτερη προτεραιότητα. Εμείς έχουμε μία επιλογή. Να επενδύσουμε στη χτεσινή Ευρώπη, την παλιά Ευρώπη ή να επενδύσουμε στο μέλλον, στο αύριο. Και τα κανάλια τα αυριανά λένε το εξή. Στο το 2050 θα, αυξηθεί, θα αυξηθούν οι ευρωπαϊκές μεταφορές κατά 80%, ε, οι επιβάτες, επιβατικές μεταφορές 50% και εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τους σιδηροδρόμους πώς θα προκριθούμε σε αυτή την τεράστια αύξηση. Δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο αν δεν επικεντρωθούμε στο μέλλον, σε αυριανές ανάγκες. Και σε αυτό που είπατε, ότι υπάρχει και κόσμος πέραν του Βερολίνου, αυτός είναι ο στόχος της επόμενης συζήτησης. Δηλαδή, έξυπνη διαδικτύωση, ε, έξυπνη δικτύωση, συγγνώμη, ε, συνδυασμένες μεταφορές και ε, τελικά οι άξονες μέσω των ο, ο, θαλασσίων οδών θα ξεκινούν από τη Σκανδιναβία και θα καταλήγουν στη Μάλτα η τελική μου απάντηση ποιος είναι ο συντονιστής για αυτά, ε, ποιος είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος του είναι καθορισμένος. Δεν είναι ότι ε, ε, ο ρόλος του είναι να συνδέσει τους, τον κόσμο, να συνδέσει τους λαούς και να μπορέσει να μεταδώσει την ουσία του έργου. Δεν είναι μεσολαβητής, ούτε είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως μόνο στόχο έχει να αναπτύξει τις συνδυασμένες μεταφορές. Είναι ο, ο είναι το, το, το λάδι το οποίο κινεί, το, το, το καύσιμο το οποίο κινεί τις μεταφορές. Είναι το, το λάδι το οποίο κινεί τον τροχό. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τα πράγματα ε, το οποίο δίνει το έναυσμα να ξεκινήσουν τα, τα έργα. Ο, όταν χρειαζόμαστε χρηματοδότηση θα πρέπει να σκεφτούμε βεβαίως την ευρωπαϊκή... Leverage to say, but if you want my money, you do it differently tomorrow. And if we don't... Ερεσιμότητα και το, το ποσοστό της μόχλευσης το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να ξεπεράσουμε την αδράνεια. Ε, υπενδύουμε στο αύριο ή διευκολύνουμε την αδράνεια. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε και τη διαμόρφωση των όρων και των συνθήκων εκείνων που θα μας επιτρέψουν την ανάπτυξη του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόξ. Να περάσω τώρα στον κύριο Σέκη, είναι ο συντονιστής για τα έργα 3 και 19. Κύριε Σέκη, έχετε 10 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προετοίμασα μερικές διαφάνειες ε, για να συνοδέψω την παρουσίασή μου, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο που σας διανεμήθηκε έγκαιρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα η πρόοδος και τη, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση με αυτά τα δύο έργα προτεραιότητας. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το PP3 αποτελεί αφορά τη σύνδεση μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας και το PP19 αφορά τη διαλειτουργικότητα στην Ιβρυκή Χερσόνησο. Τι βλέπετε σε αυτό το χάρτη όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πρώτα απ' όλα κατά το τελευταίο έτος ε, πάνω από 550 χιλιόμετρα νέων κατασκευών έχουν ξεκινήσει παρά την κρίση. Μπορείτε να τα δείτε σε αυτό το χάρτη, αν είναι αρκετά καθαρό, το κομμάτι Tour Bordeaux που αποτελεί το μεγαλύτερο ε, σιδηροδρομικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στα δεξιά το κομμάτι Νίμον Πελιέ που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι που θα επιτρέψει στο μέλλον τον Απρίλιο, από τον Απρίλιο και μετά τη σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης, Βαρκελόνης, Λιών και Παρίσιου και εκεί υπάρχει κάποια συμφόρηση και ε, η γραμμή στην Ισπανική χώρα των Βάσκων. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι με την κατάσταση παρά τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες. Όσον αφορά το PP19, καταφέραμε να δούμε νέες γραμμές προς το Αλικάντε, προς τη Γαλλική πρόσβαση προς τον Ατλαντικό, που θα συνοψίσω συνοπτικά. Πάνω από 100 χιλιόμετρα νέων γραμμές έχουν τεθεί σε λειτουργία στη περιοχή της Γαλλικίας και στη Χιρόνα. Νέα λειτουργία υψηλής ταχύτητας από Γαλλία προς Ισπανία, από τη Βαρκελόνη προς το Βορρά. Θα ξεκινήσει και θα έχει αναπτυχθεί πλήρως τον Απρίλιο του 2013. Σε μερικούς μήνες δηλαδή από τώρα. Ήδη ωστόσο λειτουργεί προσωρινά. Και αυτό θα αποτελεί τεράστιο επίτευγμα για τον ευρύτερο σχεδιασμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, διότι ξεπερνά ιστορικά εμπόδια μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Γαλλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Ταυτόχρονα η εμπορευματική σύνδεση μεταξύ του λιμανιού της Βαρκελόνης και της Γαλλίας ε, έχει τεθεί σε λειτουργία και αυξάνεται οι υποδομές βελτιώνονται και πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν και θα υλοποιηθούν νέα σχέδια κατά την επόμενη κλίση για διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που θα παρουσιαστεί μεθαύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο κατέστη δυνατό να επανεκκινήσουμε επιτυχώς τη σύνδεση προς την Πορτογαλία. την οποία έχω επισημάνει με πράσινο, δεν ξέρω αν είναι ορατή, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πορτογαλία και η Ισπανία συμφώνησαν σε μια προσέγγιση κατά φάση σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο που επρόκειται να εγκαταλειφθεί. Αυτή η προσέγγιση σε φάσεις είναι Συμβατεί με τους σημερινούς οικονομικούς και χρηματοδοτικούς περιορισμούς και θα επιτρέψει να υπερβούμε, να ξεπεράσουμε τα κενά ουσιαστικά προς την Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη από την Πορτογαλία μέχρι το 2018-2019. Καταγράψαμε επίσης πρόοδους, επίσης όσον αφορά την πιο ευρεία χρήση του η RTMS επίπεδου 2. Αυτό λειτουργεί ήδη μεταξύ Βαρκελόνης και Μαδρίτης. Και στην Ισπανία το σιδηροδρομοί υψηλή ταχύτητα αύξησαν το μερίδιο αγορά του και περαιτέρω χωρητικότητα είναι δυνατή, έχει αγοραστεί και θα συνεχιστεί μέσα στο επόμενο έτος. Φυσικά σε αυτές τις εποχές που χαρακτηρίζονται από οικονομικά προβλήματα και με το σχεδιασμό που επικοινωνούμε για το 2014-2020 προσπαθήσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο ζήτημα κλειδί της χρηματοδότησης. Αυτό το ζήτημα συζητείται πάντα το συζητήσαμε στην τελευταία συζήτηση και επιτρέψτε μου να εστιαστώ λίγο σε αυτό. Όπω γνωρίζετε, ίσω θυμάστε, πριν από περίπου δύο χρόνια μου ζητήθηκε να προεδρεύσω μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση ενός τέντη και αποφασίστηκε λοιπόν να επανεκκληθεί αυτή η ομάδα και ουσιαστικά έλαβε χώρα μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη. Σκοπός ήταν να επιχειρήσουμε να αναγνωρίσουμε τα τρέχοντα σημεία συμφόρησης, τα οποία δεν επιτρέπουν την καλύτερη, τον καλύτερο συντανισμό μεταξύ δημοσίων κονδυλίων που είναι διαθέσιμα σε ευρω... επίπεδο και εθνικών κονδυλίων με ιδιαίτερη επικέντρωση στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ειδικότερα για το ζήτημα των ε, ε, εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Και αυτό που τελείωσε κομμάτι της συζήτησης που έλαβε χώρα στις διάφορες ευκαιρίες που είχαμε και ειδικότερα υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σε μια σύνοδο που οργανώθηκε από τη Δανική Προεδρία. Φυσικά εστιάσαμε την προσοχή μας σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων και στην πρωτοβουλία ομολόγων έργων. Γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει η πειραματική φάση. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτό το στάδιο, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, τι ελλείψεις αναγνωρίζονται από τους ενδιαφερόμενους του ιδιωτικού τομέα και ούτω καθεξής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, επισημανθήκε ότι το, ανώτατη, το ανώτατο ποσοστό του 20% που επιτρέπεται για τα ομόλογα έργων στο συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο αποτελεί πολύ αυστηρό περιορισμό και αυτό το ζήτημα έχει επισημανθεί ήδη στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Με πολύ ρεαλιστικό τρόπο λοιπόν προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε και εμείς και σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Τώρα για να επανέλθω στο PP3 έχουμε φυσικά το πλέον έκτημα ότι μπορούμε να αντιλήσουμε από την εμπειρία τριών πολύ σημαντικών στιτ Τουρμπορντό, Περμπινιάν Φιγέρες που ήδη χρησιμοποιείται και την οποία επισκεφθήκαμε πέρυσι από μέλη αυτής της Επιτροπής και, και η παρακαμψή Μομπελιέ. Σκόπευμε λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και του χρόνου επί του θέματος ώστε να προσδιορίσουμε πιθανούς τρόπους ώστε και αφού εγκριθεί το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλα τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ορισμένη συγκατάσταση συζήτησή μας. Ε, φυσικά μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό έργο μεγάλης εμβέλειας ε, με τεράστια ωφέλη. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε έργα πιο ελκυστικά για επενδύσεις. Για το ίδιο είδους επενδύσεις ε, σκεφτόμαστε καλύτερα έργα, πιο σαφή, πιο ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές, ε, να μπορούμε να επισημάνουμε καλύτερα τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, ωφέλη που μπορούμε να αναμένουμε από αυτά έχοντας ε, υπόψη μας τους χρήστες τη συμβολή, ιδιαίτερα, συμβολή των σιδηροδρομικών έργων σε θέματα θετικής εξωτερήκευσης, σε ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί σε πολλές συζητήσεις και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να προσδώσουμε κάποια αξία σε αυτή τη θετική συμβουλή, συμβολή των σιδηροδρόμων, των επενδύσεων σε σιδηροδρόμους και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα ώστε να συνεισφέρουμε στη λύση που θα δοθεί χρηματοδοτικά με τα διαθέσιμα μέσα και φυσικά να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες συνέργειες με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Τι θα, γίνουν με, τι θα γίνει με το PP3 και το PP19 στο εγγύς μέλλον, το PP3 θα χωριστεί στους δύο νέους διαδρόμους του Ατλαντικού και της Μεσογείου. από το Αλγεσίρας μέχρι το σύνορο με την Ουκρανία. Κοιτώντας λοιπόν συγκεκριμένα κομμάτια αυτού του διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου Λίον Τωρίνο, για το τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί κομμάτι μιας διαδρομής άνω των 5.000 χιλιόμετρων που συνδέει τον αποτρονότο της Ευρώπης ως ε, ένα σημείο όσο το δυνατόν πιο ανατολικά. Περιλαμβάνει επίσης και το διάδρομο της Μεσογείου, μια λύση κατάλληλη κατά την άποψή μου σε σχέση με το τι ζήτησε η ισπανική πλευρά εδώ και πολύ καιρό όσον αφορά τη βελτίωση στην Ισπανία. Αυτό ονομάζεται τώρα Μεσογειακός Διάδρομος, ε, κομμάτι του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Διαδρόμου, όπω βλέπετε στο χάρτη. Όσον αφορά τον Ατλαντικό Διάδρομο, φυσικά η προσωρινή λύση, προσωρινή με την έννοια ότι θα χρειαστεί να αναβαθμιστεί στο μέλλον, και θα δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας Κατά την άποψή μου έχει αργή πρόοδο. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα σε θέματα ταχύτητας περισσότερο από τη διακοπή των εργασιών στο ε, συνοριακά τμήματα μεταξύ χώρας των Βάσκων, Γαλλίας, αλλά φαίνεται σαφώς ότι η Γαλλία θα συνδεθεί έτσι καλύτερα με τη Μαδρίτη και από εκεί και πέρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τόσο τον Ατλαντικό όσο και το Μεσογειακό διάδρομο. Τα μελλοντικά έργα λοιπόν κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. σκεπτόμενος με ποιον τρόπο θα... Ποιες θα είναι οι επιδόσεις των μελλοντικών διαδρόμων το θέμα της διακυβέρνησης έχει εμφανιστεί κατά τις παλιότερες συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Διακυβέρνηση δεν σημαίνει μόνο τι θα κάνει ο συντονιστής, τι ρόλο θα διδραματίζει, προσπαθώντας να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα. Θα πρέπει επίσης όμως να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον οργανωτικό σχεδιασμό. Διότι εάν Σκοπός είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε όλο και περισσότερο μία προσέγγιση συνδυασμένων μεταφορών και να προσπαθούμε να διατηρούμε όλους τους ενδιαφερόμενους ε, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε μια οργάνωση και μια δομή αρκετά αποτελεσματική και φυσικά υπάρχει το θέμα των χρημάτων. Αναμένουμε ε, τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που θα ελπίζουμε θα εγκριθεί χωρίς μεγάλες περικοπές αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να μελετάμε και τα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα μέσα όπως τα ομόλογα Και αυτό ελπίζουμε θα μας προσφέρει νέες ιδέες ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων που ορισμού δεν επαρκούν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μιλητές η κυρία Γιάλα και ο κύριος Δεγκράντης Πασκουάλ. Μόνο 35 λεπτά έχουμε καθυστερήσει. Δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Δεγκράντης Πασκουάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Κύριε Σέκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και τα, για τα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι ήσασταν αρκετά σαφείς και ήθελα απλώς να αναφερθώ σε δύο ζητήματα τα οποία θεωρούμε ζωτική σημασίας για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Καταρχάς το θέμα των συνδυασμένων μεταφορών και της διαλειτουργικότητας. Ε, στις διαφάνειές σας ε, που αναφέρονται στην Ιβερική Χερσόνησο, η οποία είναι αυτή που ε, αφορά τους διαδρόμους που έχετε υπό τον αρμοδιότητά σας, Καταρχάς αναφερθήκατε στο ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και εκεί έχει πολύ καλή εμπειρία η Ισπανία, αξιοσημείωτη. Και από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα των διαδρομών, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε σε στενοπούς και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν για τη διαλειτουργικότητα και στους δύο τομείς να διευκρινίσετε λίγο καλύτερα ε, ε τα θέματα αυτά, γιατί γνωρίζω ότι γνωρίζετε πλήρως το ζήτημα. Επίσης, ε, και μία ερώτηση, χωρίς να σας κάνω καμία επίκριση, θέλω απλώς μια διαπίστωση από πλευρά σας. Σε ποιο βαθμό ο χρόνος εκτέλεσης μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας τόσο στον ε, διάδρομο του Ατλαντικού όσο και αυτόν της Μεσογείας ε, έχουν ε, ταύτιση, είναι ίδιος ο ρυθμός, είναι ο ένας πίσω σε σχέση με τον άλλον. τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Διότι αυτά τα πράγματα είναι ανησυχητικά. δεν σας κάνω καμία επίκριση, απλώς ήθελα να ξέρω πού βρίσκονται τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να ήμουν σαφής και σύντομος. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σέκη για την παρέμβασή του και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κύριε Σέκη, στην εικόνα που μας δώσατε είχαμε σαφώς χαραγμένους τους δύο διαδρόμους, αυτόν που περνά από την Πορτογαλία και τον διάδρομο της Μεσογείου που φαίνεται να ανησυχεί να περνάει από τη Μαδρίτη κυρίως. Δεν είδαμε όμως τι γίνεται από την Ταραγκόνα προς τα κάτω, προς τη Βαλένθια, προς τον Νότο, όπου από ό,τι γνωρίζω υπήρχαν παρεμβάσεις που είχαν σχέση με τη διαλειτουργικότητα. Υπήρξαν βελτίωση του νέου ε, διαδρόμου της, ε, της Μεσογείου και ήταν σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπήρχαν βελτιώσει από τότε που αναλάβατε εσεί καθήκοντα συντονιστή. Αν έγιναν βελτιώσει από την περιοχή τη Ταραγώνα μέχρι τη Βαλένθια. Ε, γιατί εκεί θεωρώ ότι υπήρχε εξυγχρονισμό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, στο επόμενο διάστημα, 2014-2020, το τμήμα υψηλών ταχυτώτων ε, Λισαβόνα Μαδρίτης έχει σταματήσει ή υπάρχει ελπίδα να ανανεωθεί. Διότι η Πορτογαλία από ό,τι φαίνεται αποφάσισε να προχωρήσει τις δε μεταφορές ε, πάνω από τη Μαδρίτη, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε και τι γίνεται με τον παλιό διάδρομο και αν υπάρχουν κάποιες προσδοκίες. Επίσης, για το πρόγραμμα προτεραιότητας 16, Ξέρω ότι δεν ήσασταν εσείς ε, συντονιστής του πρόγραμματος προτεραιότητας 16, ε, αλλά είχατε την εντολή ή τουλάχιστον την ε, ε, σύσταση να ενημερώσετε τον Επίτροπο για το θέμα αυτό. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει επιτευχθεί στο τελευταίο διάστημα, διότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσον στο μέλλον μπορούμε τουλάχιστον να ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν οι μελέτες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση ε, γιατί έτσι την αποκαλούμε σε άλλα θέματα. Και επίση, επειδή είστε πανεπιστημιακό, θα ήθελα να σα ρωτήσω, όταν αναφέρεστε στη συγκέντρωση, πώ θα αναλέτε το γεγονό ότι από το 2013, από τα 8, 800 εκατομμύρια προγραμμάτων, πρέπει ακόμα να δοθούν. Ε, συγγνώμη, από τα 8 δις προγραμμάτων πρέπει ακόμα να δοθούν ένα δις. Κάποιοι θεωρούν ότι το να επενδύσουν μερικά εκατομμύρια για την κεντρική διαδρομή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πιο προηγμένα συστήματα. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Σέκη για τις εξηγήσεις που έδωσε. Θα κάνω και εγώ μια προσπάθεια για να ε, προσπαθήσω να σας ρωτήσω τηλεγραφικά κάποια σημεία. Είπατε και αυτό το ακούμε σταθερά από όλους τους συντονιστές ότι είναι σημαντικά τα συνοριακά τμήματα. Ε, στην γραμμή προτεραιότητας 3 για το τμήμα του Ατλαντικού όπου ε, διασχίζουμε την ε, περιοχή της Ιβηρικής υπάρχει πρόβλημα στα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Θα ήθελα να γνωρίζω με όλες τις τεφλονικές που υπήρχαν αν υπάρχει κάτι για τη θέση της γαλλικής κυβέρνησης και αν υπάρχει κάποια συμφωνία για να προχωρήσει το τμήμα αυτό μεταξύ γαλλικής και ισπανικής κυβέρνησης. Επίσης, ανεφεθήκατε σε διάφορα χρηματοδοτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα προτεραιότητας και θα ήθελα να σας ρωτήσω λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια πολύ κακή οικονομική κατάσταση και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το Connecting Europe σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά η Ισπανική κυβέρνηση μείωσε κατά 40% τα προγράμματα υποδομών της, αν γνωρίζετε, αν θα προχωρήσει η γραμμή ε, η οποία είναι γνωστή ως ε, Y πασκα η Μπάσκα, η γραμμή της χώρας των Βάσκων και αν θα υπάρξει κάποια διακοπή στη γραμμή αυτή. Επίσης, Θεωρείτε ότι το να εντάξουμε νέα προγράμματα μπορούν να ε, θέσουν κινδύνο τα προγράμματα τα οποία έχουμε ήδη εξελίξει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ. Ε, Μαδρίτη Λισαβόνα. Μεταξύ Κατφέρες και Μπάγια σε ένα μικρό τμήμα, έχουν ξεκινήσει εργασίες είναι η ευρωπαϊκή κανονική γραμμή, γιατί είναι φαρδιά γραμμή. Πώς ρυθμίζεται αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι η Ισπανία επέλεξε την κανονική διάσταση των γραμμών. Δεύτερον, όσον αφορά τα θετικά εξωτερικά, τα θετικά εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν το έργο. Ποια είναι αυτά. Και τρίτον, η άμεση διασύνδεση ε, από τη Γαλλία στα σύνορα. Η μία διαδρομή θα είναι έτοιμη το 2020. Όλα έχουν σημειωθεί με κόκκινο και προς τη Μεσόγειο το 2020. Είσαστε αισιόδοξο για αυτό τον άξονα, ε, για τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία έχει οικονομικά προβλήματα και αν το τμήμα Λιόν-Τωρίνο είναι πιο σημαντικό, τότε αυτές τις δύο γραμμές προς Νότον δεν θα μπορέσετε να τις χρηματοδοτήσετε. Ο κύριος Σέτσι. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Να απαντήσω εν συντομία όλα αυτά τα σημαντικά ερωτήματα. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσα διμερώς να διευκρινίσω κάποια πράγματα, αν δεν είναι αρκετά σαφής. Διαλειτουργικότητα. Η Ισπανία, κατά την άποψή μου, είχε αξιοσημείωτες επιδόσεις, παρά τις δυσκολίες ε, και τη διαφορά στο άνοιγμα των ε, τροχών, στο εύρος των τροχών και το καθεξής. Το δίκτυο υψηλή ταχύτητα βέβαια είναι στις ευρωπαϊκές διαστάσεις του ανοίγματο των τροχών, αλλά από εκεί και πέρα ε, το περαιτέρω τμήμα του σιδηροδρόμου ε, αρχίζει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και αυτό φυσικά επιτρέπει να χρησιμοποιούν και να συνεπάρχουν και το άνοιγμα των τροχών της Ιβυρικής Χερσονήσου και το άνοιγμα των ευρωπαϊκών διαστάσεων. Ε, υπάρχει λοιπόν και οι φυστάμενες πιο σημαντικές γραμμές αναπτύσσονται και ε, υπάρχει συνέπεια κατά αυτόν τον τρόπο. Το ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, είναι πολύ καλά εφαρμοσμένο στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου και σε αυτό το τμήμα η Ισπανία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά το χειρισμό και τη σηματοδότηση και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση ε, για λόγους ε, βέβαια ε, χρόνου χρειάστηκε να είμαι πολύ συνοπτικό στην παρουσίασή μου, γι' αυτό και δεν σας τα είπα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ποσοστό και ο ρυθμός εκτέλεσης. Δύσκολο ερώτημα. Υπάρχουν διαφορές ως προς τα χρονοδιαγράμματα, αλλά βεβαίως ε, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, ε, πότε εγκρίνεται ένα σχέδιο, τι γίνεται με την τοπική κοινότητα, ε, το γαλλικό σύστημα και ούτω καθεξής. Τα πάντα λοιπόν κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξο ε, και για να απαντήσω και στην ερώτηση του κυρίου Κράμερ, θεωρώ ότι για το τμήμα της Μεσογείου, όχι μόνο θα έχουμε τη νέα γραμμή εν πλήρη λειτουργία ε, μέχρι τον επόμενο Απρίλιο, αλλά η στενοπός που βρίσκεται στο Μομπελιέ ε, θα επιληφθεί, θα ληφθεί απόφαση και θα διορθωθεί και το πρόβλημα αυτό. Δεν ε, θεωρώ ότι αυτό είναι εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλο πρόγραμμα. Πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος ε, Μπρινκχόρστ προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση θα βρει την απαραίτητη χρηματοδότηση για όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν προτεραιότητα. Και κυρίως ε, οι πλέον αρμόδιοι θα συμμετέχουν ε, με επιτυχή τρόπο, θα υπάρξει σύμπρεξη και με τον ιδιωτικό τομέα, όπως έγινε και για το τμήμα του Μπορντό. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν. Ο διάδρομος της Μεσογείου Κυρία Γιάλα Σέντερ, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι συνάδελφοί σας, ότι το τμήμα Ταραγκώνα Βαλένθια βελτιώνεται και στο νέο σχεδιασμό ο διάδρομος θα πηγαίνει μέχρι το Λιγιζέιρας. Δεν θα είναι πλήρως λειτουργικός, δεν θα πηγαίνει από όλη την ακτή, αλλά ε, θεωρώ ότι υπάρχει ε, περιθώριο για βελτίωση προς τον, νόσο και να βρεθούν, ε, προς τον νότο συγγνώμη, και να βρεθούν και λύσεις οι οποίες είναι συμβατές με τις περιβαλλοντικές, ε, κλπ. απαιτήσεις. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει πρόοδος και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το κομμάτι Λισαβόνα Μαδρίτη, η λύση η οποία προτείνεται και ε, επί της οποίας συμφώνησαν και οι δύο κυβερνήσεις είναι ε, μια λύση που είναι κατά τη διαφορετική από την προηγούμενη πρόταση, να υπάρχει μια πλήρως ε, λειτουργούσα γραμμή υψηλής ταχύτητας ε, μεταξύ Λισαβόνας και Μαδρίτης. Θα έχουμε δύο διαδρόμους, έναν της Ιβηρικής και έναν με, ευρωπαϊκές, με ισπανικές και έναν με ευρωπαϊκές διαστάσεις εύρους τροχών και θα έχουμε διαχείριση της κίνησης μεταξύ Λισαβόνας και Μαδρίτης. Θα εξοικονομείται αρκετός χρόνος και ε, θα αιτιολογείται έτσι και η επένδυση από ισπανικής πλευράς. Ιδάλω θα φτάνουμε στα σύνορα και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να προχωρήσουν. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα επιτρέπεται και η μεταφορά εμπεροβμάτων. Θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω από τους πορτογαλικούς λιμένες που βρίσκονται σε πολύ ευνοϊκή γεωγραφική θέση, διότι είναι οι λιμένες οι οποίες είναι πιο κοντά προς το δυτικό τμήμα της διαδρομής, που είναι πιο κοντά στη νέα διορίγμα του Παναμά και ούτε καθαξής. Εάν όμως δεν συνδεθεί ε, τουλάχιστον με μία διαδρομή διπλής χρήσης και ευρωπαϊκών και ισπανικών ε, διαστάσεων, όλα ε, θα καθυστερήσουν φυσικά. Τι αποφασίστηκε λοιπόν και τι κατά την άποψή μου θα υλοποιηθεί εγκαίρως είναι ε, το τμήμα το οποίο βλέπετε στο χάρτη που είναι στο πιο νότιο τμήμα. Ε, είναι εν μέρει ανύπαρκτο και υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλες βελτιώσεις, αλλά υπάρχει ε, η χαρτογράφηση και μέσω αυτής της συμφωνίας υπήρχε η δυνατότητα να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή, τα χρήματα από, την, ε, ε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα και θεωρώ ότι για την Πορτογαλία αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό διότι το ήθελαν και εν ώψη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Τέλος, η σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών της χώρας των Βάσκων και την, του Ισπανικού και του Γαλλικού τμήματος. Από την Ισπανική πλευρά δίνεται εντύπωση ότι τα πάντα προχωρούσαν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνεται και πρόοδος και από την άλλη πλευρά. Και νομίζω ότι γρήγορα θα υπάρχει βελτίωση τουλάχιστον της υφιστάμενης κατάστασης. Και για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές τη σπάση ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό οδικής κυκλοφορίας από τα βόρεια σύνορα της Ισπανίας και, τη, και στην Πορτογαλία χρειάζεται μια άλλη λύση που να είναι και περιβαλλοντικά συμβατή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο εξακολουθούμε να πιέζουμε ε, όλες τις ε, ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και σκοπεύω να επικεντρωθώ στο μέλλον σε αυτό το τμήμα και ελπίζω να μπορέσω να σας αναφέρω κάποιες θετικές εξελίξεις και για τις δύο πλευρές του προγράμματος προτεραιότητας 3. Ε, Βέβαια, περισσότερη προσοχή ε, χρειαζόμαστε ίσως την ε, άλλη σύνδεση, η οποία ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα εγγένεια. Περνάμε τώρα στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων με τον συνάδελφο κύριο Σαβαρή για το έργο προτεραιότητας 22. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας ενημερώσω λοιπόν για την κατάσταση του PP22. E Les problèmes d'interopérabilité. Προβλήματα διαλειτουργικότητας αντιμετωπίζουμε όπως βλέπετε. C'est moi qui le, c'est moi qui le manipule Chacun là Oui, mes chers collègues, il s'agit donc de... Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε λοιπόν για ένα σιδηροδρομικό έργο, όπως γνωρίζετε, μήκους 3.793 ε, χιλιόμετρων που αποτελεί μία πύλη εισόδου από την Ανατολή προς τη Δύση και που αποτελείται από πολύ παλιά ιστορικά δίκτυα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους όσον αφορά τα πρότυπα. Στόχος ε, είναι η δημιουργία δύο ηλεκτροδοτούμενων γραμμών ERTMS 22 τόνων ε, υποστήριξη στο σύνολο της γραμμή. Υπάρχουν τρει κλάδοι προ τα Ανατολικά, μία προ τη Βρέστη, προ την Ρεμβέργη και προ το Βερολίνο από την Πράγα. Και όπω βλέπετε τρέχει την Αυστρία, την Ουγγαρία προ την Κωνσταντζα και τον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα προτεραιότητα που ψήφισε στη λίστα Βενμίρτ και που σήμερα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Ποιες ήταν λοιπόν οι κύριες πρόοδοι φέτος τα εξή υλοποιήθηκαν. Με κόκκινο βλέπετε αυτά που δεν έχουν υλοποιηθεί και με πράσινο αυτά που έχουν πρακτικά ολοκληρωθεί. Στην δημοκρατία της Τσεχίας μέχρι τα γερμανικά σύνορα οι δύο κλάδοι είναι πλέον συμμορφούμενοι με τις προδιαγραφές. Αντιθέτως η γραμμή προς τον νότο η οποία ωστόσο δεν θα μπορέσει να τρέξει με 140 χιλιόμετρα που πηγαίνει προς τον Ίσ, διότι περνάει μέσα από βουνά, είναι μία γραμμή, ουσιαστικά ειδικά για εμπορεύματα. Μετά έχουμε το σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, μια πανέμορφη, ένα πανέμορφο νέο σιδηροδρομικό σταθμό που σας καλώ να επισκεφθείτε, διότι αποτελεί άριστο παράδειγμα συνδυασμένων μεταφορών αστικών και μεγάλων αποστάσεων και πρόκειται για, μια, για ένα παλιό σταθμό από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και που αποτελεί κομβικό σταθμό αυτή τη στιγμή στρατηγικό για την Αυστρία μεταξύ Ανατολή Δύση και Βορανότου, ουσιαστικά κομβικό σημείο από τη Βαλτική προ το Μεσόγειο, από τον Εύξενο Πόντο προ τη Βαλτική. Δεν, έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τεθεί ακόμα πλήρω σε λειτουργία, αλλά έχει ολοκληρωθεί. Για την Ουγγαρία η οποία έχει ένα δίκτυο σχεδόν ολοκληρωμένο. Ακόμα υπάρχει το κομμάτι προς την Αυστρία που χρειάζεται βελτίωση. Ουσιαστικά οι εργασίες ε, εστιάστηκαν στο Μπέκε Σαμπάλε και στο Κοσασά κάποια χιλιόμετρα από τα ε, ρουμανικά σύνορα. Βρίσκονται σε τελική φάση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρω σταματάνε στο Κοσάσα, παραμένουν, απομένουν μερικά χιλιόμετρα μίας μονογραμμή που θα αποτελέσουν προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες. Στη Ρουμανία πολύ μεγάλα τα έργα, αλλά αυτός ο άξονας Κωνσταντζας Βουκουρέστη έχει λάβει προτεραιότητα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έχουν ανατραπεί λίγο οι προτεραιότητες ευρωπαϊκές με γρήγορο ρυθμό αυτό το κομμάτι και στα ουγγρικά σύνορα όπου γίνονται τεράστιε προσπάθειε από του Ρουμάνου μεταξύ του Αράτ και του Κοτιτσί που βρίσκεται στα σύνορα. Οι Ουγγροί λοιπόν έχουν καθυστερήσει λίγο στη δική του πλευρά. Μεγάλες εξελίξεις των άξων βορρα βορρά-νότου θα είναι η ολοκλήρωση της γέφυρας στο Δούναβη. Ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 4-5 μήνες. Βλέπετε εδώ το, η γέφυρα Βίντιν Καλαφάτ τον 19ο αιώνα βομβάρδιζαν ή μία ακτή την άλλη. Ήταν ένα σημείο επαφής. Υπάρχει επίση και άλλη μια γέφυρα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας που ονομάζεται Ρούσε. Αυτή η, Γερμανία, αυτή η γέφυρα θα χρησιμοποιείται τόσο επαφη οδικές όσο και αλλη μια γεφυρα μεταξυ βουλγαριας και ρουμανιας που ονομαζεται αυτη η γερμανια μεταφορές. Και σε λίγο ναι, αυτό, αυτή θα είναι, αυτό θα είναι το μεγάλο γεγονό του έτου και βλέπετε ωστόσο το κόκκινο κομμάτι που παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Δεν είμαι καθόλου βεβαίω κατά πόσο θα μπορέσει να προοδεύσει. Διότι πολύ λογικά η Βουλγαρία όπως και η Ρουμανία δίνουν προτεραιότητα στα κομμάτια από την Ανατολή προς τη Δύση. Οι Βούλγαροι κάνουν προσπάθειες προς τον Ευξενοπόντο, στο λιμάνι του Μπουργκάς, και σήμερα εστιαζούν επίσης τις προσπάθειές τους ε, σε ένα κομμάτι που θα ανήκει στον επόμενο διάδρομο. Η Κομισιόν λοιπόν καλά έκανε και ενσωμάτωσε αυτές τις νέες προτεραιότητες προς την Τουρκία και που θα αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα σε αυτή την περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται μια σύρακα ε, υποθαλάσσια στο Βόσπορο από τους Τούρκους. Εκεί θα έχουμε λοιπόν ανατροπή τορών Μεγάλες αλλαγές λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, το κόκκινο από το βορρά προς το νότο, αλλά εκεί ουσιαστικά έχουμε αδιέξοδο προς την Ελλάδα, όπου έχουν γίνει έργα παρότι αντιμετωπίζει η Ελλάδα σημαντικές δυσκολίες, ε, για τις οποίες θα σας μιλήσω αργότερα, αλλά ουσιαστικά καταλήγουμε σε αδιέξοδο βορρά της Ελλάδας, διότι μιλάμε για μια γραμμή μονή, που πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα το πολύ σε εξαιρετικά στενά φαράγγια όπου κανείς δεν προβλέπει εκτός αν υπάρξουν πολλά κονδύλια να διευρυνθούν τα φαράγγια αυτά και έτσι πια δεν υπάρχουν πλέον επιβατικές ε, μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Σόφιας. Υπάρχουν κάποιες λίγες μεταφορές εμπορευματικές. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση σε αυτή τη γραμμή αυτά που έχουν γίνει το 2011-2012. Μπορείτε να δείτε σε αυτό το γράφημα, σε αυτή τη γραφική παράσταση, ότι ουσιαστικά το κομματικό στάντζα το βλέπετε με πράσινο, αυτά που βλέπετε με κόκκινα δεν έχουν υλοποιηθεί, αυτά που βλέπετε με πράσινο έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Όπως βλέπετε ε, έχουν σημαντικές πρόοδοι στο ανατολικό κομμάτι προς την Κωνσταντζα, προς τον Μπουργκάς. Ελάχιστη πρόοδος, ε, όπως βλέπετε στην κόκκινη γραμμή κάτω, στο κομμάτι από το Αράντ, στη Ρουμανία, στα σύνορα με την Ουγγαρία, χρήτα ελληνικά σύνορα με τη Βουλγαρία. Πρόβλημα λοιπόν στον άξονα βορρανό του, μεγάλε πρόοδοι από τη Δύση προ την Ανατολή σαν έναν ανταγωνισμό υπέρ τη μαύρη Θάλασσα, που μου φαίνεται λογικό. Αυτέ οι δύο χώρε προσπαθούν να εστιαστούν στην κίνηση με την, προς την Κεντρική Ασία με τώρα την κυκλοφορία κάτω από το Βόσπορο που θα επέλθει και που αλλάζει τη γεωγραφία ουσιαστικά κάπω. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους Τούρκους γιατί θα αποτελεί μια μόνιμη σύνδεση θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα ως κατεπήγον. Τώρα, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικά υποσύνολα. Βορειοδυτικά έχουμε τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία που εργάζονται διμερώς αρκετά σωστά. Με ωστόσο μία δυσκολία που πρέπει να σας αναφέρω, διότι τη συνάντησα, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα, ως προτεραιότητα την ανακαίνιση του κλασικού της δικτύου παρά να επενδύσει σε νέες γραμμές. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για, την, για τη Δρέσδη, όπου οι Τσέχοι και οι Σάξονες σχεδιάζουν μια μελέτη για μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ Δρέσδης και Πράγας, ενώ η Γερμανία δίνει προτεραιότητα περισσότερο στο κομμάτι από το βορρά προς τον νότο, παρά στο κομμάτι από τη Δύση προς την Ανατολή. Οι Τσέχοι λοιπόν βρισκόνται απομονωμένοι, διότι αυτή τη στιγμή δεν ε, υπάρχει γερμανική προτεραιότητα, δεν αποτελεί αδιαφορία για τη σύνδεση της Πράγας τόσο με την Ερεμβέργη, με έργα στο γερμανικό κομμάτι, αλλά και με τη Δρέσδη και πέραν αυτής. Η Κομισιόν, όπως γνωρίζετε, στο μελλοντικό διάδρομο έχει συμπεριλάβει το Ρόστοκ, μιλήσαμε πολύ γι' αυτό, και το Αμβούργο. Και ελπίζουμε ότι οι Γερμανοί θα θεωρήσουν ότι η Πράγα και η ενδοχώρα των λιμένων τους ε, αξίζουν την προσπάθεια για να γίνει αυτός ο άξονας βορρανο Ανατολής. Νοτιοανατολικά έχουμε υλοποιήσει αυτό που ίσως αποτελέσει πλατφόρμα διακυβέρνησης ενός διαδρόμου διότι εγώ, αφού το ζήτησαν τα κράτη-μέλη, προεδρεύω τακτικά συνεδριάσεις ε, στις οποίες συμμετέχουν τα τέσσερα Υπουργεία Μεταφορών των τεσσάρων χωρών, συμμετέχουν οι ιστορικές ε, συνδρομικές εταιρείες, οι διαχειριστές υποδομών των τεσσάρων χωρών είναι παρόντες. Αυτός είναι ο συντονισμός μεταξύ αυτών των τεσσάρων χωρών. Και ε, μετά εμείς οι Ευρωπαίοι ε, συντονιζόμαστε μεταξύ μας. Είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα και τέσσερις γενικές διευθύνσεις και τώρα συζητάμε τη διαχείριση του διαδρόμου, εμπορευματικού διαδρόμου αριθμού 7. Τι κάνουμε σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ε, προσπαθούμε να βολιδοσκοπήσουμε τις επιθυμίες του και τις προθέσεις του κάθε κράτους μέλους. Αλλά ουσιαστικά προχωράμε με δύο τρόπου. Υπάρχουν δύο λειτουργικότητε σε αυτή την πλατφόρμα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε κάνει μελέτε. Μελέτε στο σύνολο αποτελούν πολύτιμο στοιχείο για το σύνολο του έργου προτεραιότητας. Ανά πάσα στιγμή, για κάθε χιλιόμετρο, γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση του δικτύου. Δεύτερο κομμάτι, κοινωνικο-οικονομικές ε, πτυχές, ανάλυση, πλεονεκτήματα που μας δείχνουν ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε ορισμένα κομμάτια, τα οποία ενδεχομένω δεν είναι τα πιο ακριβά, αλλά θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα και αυτό προσθέτει αξία και για τα τέσσερα υπουργεία των τεσσάρων κρατών μελών. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργικά είμαστε καλά οργανωμένοι όσον αφορά τι εργασίε, πολύ λιγότερο όσον αφορά τι οικονομικέ μελέτε και τι μελέτε επιπτώσεων. Με αυτέ τι μελέτε τροφοδοτούμε τι στρατηγικέ των διαφορών υπουργείων. λαμβάνοντα υπόψη τι πληροφορίε των δικτύων και τι προβλέψει κυκλοφορία. Αλλά ουσιαστικά εδώ κατακαιρματίζουμε κάπως το έργο αυτό σε μικρά κομμάτια με τα επιμέρους ωφέλη τους. Και από την άλλη ζητάμε από τα κράτη-μέλη ένα προγραμματισμό και επενδύσεις εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Στην επόμενη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα στην Αθήνα θα ξεκινήσουμε. Τους ζήτησα να μου, να δώσουν ένα προγραμματισμό για την επόμενη δημοσιονομικές προοπτικές ώστε να δούμε τι είναι εφικτό και τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτά τα κράτη-μέλη. Εντάξαμε λοιπόν το διάδρομο. Τι παρατηρήσαμε. Παρατηρήσαμε και τα διασυνοριακά κομμάτια. Εκεί λοιπόν ε, μας εκπλήσει το εξής γεγονός. Οι τεράστιες δυσκολίες μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας δεν οφείλονται σε μη συντονισμό μεταξύ Ούγγρων και Ρουμάνων, συνεργάζονται άριστα μεταξύ του. Έχουν μάλιστα μία μεικτή ομάδα στο κουτί, στη Ρουμανία. 12 ώρες αναμονής για ορισμένα τρένα, ειδικά τρένα εμπορευμάτων. Σέγγεν. Και είναι δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Γίνονται προσπάθειες από την Ουγγαρία, ειδικότερα. Έχουμε επισημάνει σαφώς το πρόβλημα. Μίλησε για τις μελέτες. Τώρα θα προχωρήσω πιο γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος. Τα συμπεράσματα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα που θα σα πω θα είναι λίγο προσωπικά δικά μου. Το πρώτο είναι ότι οι επιπτώσει τη κρίση των δημοσίων προπολογισμών γίνονται αισθητέ και αυτό που ζητάμε εμεί από τα κράτη-μέλη είναι πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή, αντί να αξιολογούν και να λειτουργούν το σύστημα σε μεγάλα κομμάτια, να έχουν μια προσέγγιση με μικρά βήματα, με επενδύσεις ίσως λίγο πιο μετριοπαθείς, αλλά που παράγουν άμεσα αποτελέσματα. Επιδιώκουμε λοιπόν διαρκείς πρόοδους, αλλά που ενίοτε εστιάζονται στη διαλειτουργικότητα, για παράδειγμα, ή στην υλοποίηση του ERTMS, ή σε κομμάτια τα οποία δεν είναι υπερβολικά ακριβά εντό εισαγωγικών. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση, μια έτσι απέτηση ρεαλισμού και επένδυση σε όριμα έργα το οποίο απαντάει και στι ανησυχίε μα για τι δυνατότητε απορρόφηση. Έχουμε λοιπόν προσδιορίσει τρει άξονε απόλυτη προτεραιότητα για του επόμενου μήνε. Τη την τεχνική διαλειτουργικότητα, ε, το ζήτημα της Βουδαπέστης ε, όπου συζητείται παράκαμψη ενδεχομένως με μια τρίτη γραμμή βάσει μιας ε, κεντρικής γέφυρας μπορεί να χρειαστεί 20 χρόνια. Και τέλο, εστίαση στα διασυνοριακά κομμάτια από τεχνική άποψη. Το Σέγγεν είναι μια άλλη ιστορία. Αναφέρθηκε ένα πρόβλημα. Αυτέ οι χώρε θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει κάπω τα υλικά. Είναι σύνθετο αυτό το θέμα. Έχει ξαναγίνει, αλλά θα επιτρέψει να προχωρήσει η διαλειτουργικότητα. Δεν, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε οποιοδήποτε υλικά σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της ανανέωσης ε, των τρένων ε, και της διαλειτουργικότητας ε, είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Εγώ πήρα ένα τρένο το οποίο ήταν του 61, λειτουργούσε πολύ καλά, πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι ακριβώς διαλειτουργικό. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που τέθηκαν. Δεύτερο, αυτό που βλέπω είναι μια γεωγραφική στρέβλωση του έργου ε, προτεραιότητες ε, προς την Τουρκία και όσον αφορά το βαλκανικό ζήτημα ουσιαστικά βρίσκονται σε διέξοδο οι Έλληνες ε, λόγω αυτού του ζητήματος της οδού προς τα κάτω. Βλέπετε ότι η οδός αυτή η μία είναι 1300 χιλιόμετρα και η άλλη 1032 και σήμερα είναι σαφώς ότι όλα τα επιβατικά τρένα που φεύγουν από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη περνάνε από τα Βαλκάνια διότι κανένα πλέον δεν περνάει από τη Σόφια η γέφυρα Βιντιν Καλαφάτ που θα είναι ένα εξαιρετικό έργο που για πολύ καιρό υπήρξε οδική γέφυρα με έλλειπη πρόσβαση. Θα πιέσουμε λοιπόν τα δύο κράτη-μέλη να αυξήσουν τις προσβάσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν έχουμε φωτογραφία, νομίζω είχαμε μία για να σας δώσουμε μια εικόνα του τι γίνεται στο Βιντιν Καλαφάτ. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Τέλος, όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών. Αυτή είναι η γραμμή που καταλήγει στη γέφυρα Βιντίν Καλαφάτη. Είδατε αυτή την καταπληκτική γέφυρα και έχετε μία μονή σιδηροδρομική γραμμή νότια της Σόφιας, ε, συγγνώμη, βόρεια της Σόφιας για πολλά χιλιόμετρα που οδηγά προς την γέφυρα Βιντίν Καλαφάτη. Δηλαδή θα έχουμε μία γέφυρα που θα είναι περισσότερο γέφυρα για αυτοκίνητα παρά για σιδηροδρόμους για πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά και τα δύο μέρη δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτή των εμπορευματικών μεταφορών. Αλλά το έργο προτεραιότητας, ε, τα κράτη-μέλη το θεωρούν όλο και περισσότερο ως ε, ένα έργο που αφορά τα εμπορεύματα. Σημαντικό λοιπόν να εντάξουμε το πρόγραμμα αυτό σε διάδρομο. Εγώ δεν βλέπω πολύ καλά ποιε είναι οι πολύ σημαντικέ οδικέ επενδύσει που γίνονται, ενώ εμεί σπρώχνουμε τι ε, συνδρομικέ επενδύσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητή αναγκαία η προσέγγιση τη Κομισιόν ώστε να κάνουμε γεωγραφία περισσότερο από μηχανολογία. Πιστεύω ότι εδώ μπορώ να ολοκληρώσω τα συμπεράσματά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κούν, Σεναλόβα, Λίχτεμπεργκερ, Κράμερ, Αγιάλα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριος Κούν, ευχαριστώ πολύ για τις δραστηριότητες του. Δεν είναι μόνο ένα δύσκολο τοπογραφικό έργο αυτό, αυτός ο άξονας 122 ε, είναι και πολιτικά δύσκολος άξονος, είναι περίπλοκα τα πολιτικά δεδομένα, δεδομένου ότι έχουμε νέα κράτη-μέλη, ε, δύσκολη κατάσταση χρηματοδότησης κλπ. Αλλά υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Γερμανίας και αυτό με συγχύζει. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξή. Έχοντας υπόψη το συνδέοντας, τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη και έχουμε καθορίσει ένα διάδρομο στον οποίο θα συμμετωθούν αυτά τα έργα προτεραιότητας. Και είπατε από την Ασίνα, Κωνσταντζα, ε, Σβάτσβαλτ, Μέλανα Δημός κλπ. Μεσοδρέσδης θα επεκταθεί αυτό το τμήμα το ίδιο προς την κατεύθυνση όπως όμως καθορίσαμε και τις κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να συνδέσουμε ε, τις βόρειες ακτές με τις νότιες ακτές. Και πέραν της ε, Δρέσδης προς το Βερολίνο και εν συνεχεία ρωστο το Καμβούργο προς της μας, είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο άξονας και έχουν ενσωματωθεί και οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, οι διπλές γρασιδρομικές γραμμές προς τη Δρέσδη και η διασταύρωση προς το Σάντο πρέπει, απαιτεί ε, bypass, παράκαμψη. Η κυρία Σαναλόβα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σαβαρή για την παρουσίασή του. Έρχομαι από την Τσεχική Δημοκρατία και θα ήθελα να σα ρωτήσω για τη σύνδεση Τσεχικής Δημοκρατίας ε, Γερμανία. Αναφέρατε διάφορε προτεραιότητε, βασί των οποίων η Γερμανία προτιμά τη σύνδεση από βορρά προς νότο. Και σε κάθε περίπτωση για μας βέβαια από την άλλη πλευρά είναι πιο σημαντική ο άξονας από δύση προ ανατολή. Και όταν μιλάμε για προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή για να ρίξουμε τελείως το σιδηρόν τείχος που παραμένει στις μεταφορές μετά από 20 χρόνια. Πιστεύω ο ρόλος των συντονιστών υπό αυτές τις περιστάσεις θα καταστεί εξαιρετικά σημαντικός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για το έργο σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Η σύνδεση μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας και Γερμανίας, όπως γνωρίζουμε, Υπάρχουν πολλά σχέδια Πράγα Νιρεμβέργη ή Πράγα Μόναχο. Ποια είναι η δική σας άποψη. Δεύτερη ερώτηση, η σύνδεση μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας και Αυστρία μεταξύ του Μπουδβάης και του Λίντς. Γνωρίζετε κατά την ανασκόπηση της ρύθμισης ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, αυτό ε, παραμελήθηκε. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η σύνδεση. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ. Και εγώ αναφέρομαι στη, στο τμήμα μεταξύ Πράγας και Βιέννης. Χαίρομαι που συμπεριλαμβάνει και ένα σημαντικό έργο, τη γραμμή Zoomer Hour, είναι ένα τμήμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό και για τις, και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό το τμήμα, διότι έχει και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, οικονομική αξία. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το, το Είχαμε κάνει μια επίσκεψη εκεί και αυτό το έργο το οποίο δεν είχε ευρεία συνένεση, είναι και πολύ ακριβό όσον αφορά το σταθμό, το συνδρομικό σταθμό στο Μπρουνό. Είχαμε μελετήσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και εν συνεχεία στα αστριακά σύνορα μεταξύ Βιέννης και Ουγγαρίας υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, ένα ενδιαφέρον τμήμα με, μεταξύ των τριών χωρών. Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία. Η κυρία Γιάλα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζήλ Σαβαρή για την παρουσίασή του. Για την πλατφόρμα συντονισμού που θα μπορούσε να αποτελέσει και πρότυπο για τους μελλοντικού μας διαδρόμους, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οι μελέτες και ο συντονισμός που γίνονται σε αυτή την πλατφόρμα με τους ε, ε, υπευθύνους, τους διαχειριστές των υποδομών, τους υπευθύνους των Υπουργείων και καθεξής. Ε, αλλάζουν εξαιτία αυτού του συντονισμού τα εθνικά σχέδια ή τα πάντα παραμένουν ε, αυστηρά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο αυτό ο συντονισμό τον εθνικό σχεδιασμό, διότι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να το συμπεριλάβουμε και τους υπόλοιπους σχεδιασμούς. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και για αυτή τη διευκρίνηση, αυτό που είχαμε στο πρόγραμμα προτεραιότητας 22, η σύνδεση μεταξύ Πράγας ε, και Lights εξαφανίζεται, δεν θα υπάρχει στο Connecting Europe. Επίσης, λέτε ότι ο διάδρομος προτεραιότητας ε, θα γίνει διάδρομος εμπορευματικό. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ενδιαφέρον για επιβάτες για να πάνε μέχρι Γερμανία, ε, από Γερμανία σε Τσεχία. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για επιβάτες, ε, αφού βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη δέσμη μέτρων ε, για τους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Κράμ. Ε, Ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Με εκπλήττουν λίγο οι Τσέχοι. 50 μεγάλα έργα και θέλουν ε, βεβαίω την Πράγα, θέλουν το, το τμήμα Δρέστη Βιέννη, θέλουν τον πλατείνουν τον Έλβα, θέλουν επίση προ την κατεύθυνση επίσης και στον Μπρνό, ε, στο να, να, να κατασκευαστεί ο σταθμός. Ε, αυτά χωρίς συγχρηματοδότηση δεν γίνεται και δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν η συγχρηματοδότηση κατά το 20% πέντε μεγάλων έργων, ας αποφασίσουν για ένα έργο. Καταλαβαίνω για τη Γερμανία ότι ο άξονα τη Ρεμβέργη Πράγας δεν είχε προτεραιότητα όταν υπήρχε το σιδηρούν προσωπείο, το ψυχρός πόλεμος, αλλά τώρα όσον, αφορά τον συνδρομικό σταθμό στο Μπρουν, και ρωτώ τον κύριο Σαβαρή, έχετε πει ότι δεν θα πάρουν ε, δεκάρα, όπως λέμε, ή δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ εάν θέλουν να αναδιαμορφώσουν το σταθμό, διότι μία αναμόρφωση ενός συνδρομικού σταθμού δεν γίνεται με ευρωπαϊκά χρήματα. Το έχετε πει αυτό ξεκάθαρα στους Τσέχους. Και ποια είναι η αντίδραση. Όσον αφορά τη γέφυρα πάνω από το Δούναβι, θα πρέπει να είναι μια συνδυασμένη γέφυρα και για αυτοκίνητα και για σιδηροδρόμους. Έχετε λάβει υπόψη τις ε, μακρινές αποστάσεις, δηλαδή τις μακρινές μεταφορές. Και τι γίνεται με αυτή τη γέφυρα. Thank you very much, Gilles. You Ευχαριστώ. Είσαι τυχερός, διότι έχουμε ε, ε, περάσει όλους τους συντονιστές και για χάρη σου αναφέραμε και τα ποδήλατα. Λοιπόν, μπορείς να απαντήσεις παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κούν, δεν θα ήθελα να ερμηνεύεται αυτό που συμβαίνει μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας ως ε, αντίθεση μεταξύ Τσέχων και Γερμανών. Το ζήτημα είναι ότι ο συντονιστής διαπιστώνει πως οι δύο χώρες δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες και οι δύο είναι σχετικά λογικοί. Οι Γερμανοί θέλουν μάλλον έναν άξονα από το Βερολίνο προ τον νότο τη Γερμανία, το Μόναχο, ω πρώτη προτεραιότητα. Δεν θέλουν να επενδύσουν σε νέε ναι, επενδύσει, Αυτά μα λένε. Όταν λέω Γερμανοί, μιλάω για το Ομοσπονδιακό κράτος. Η Σαξονία μόνη τη θα ήθελε πραγματικά να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ πράγα και δρέσδη. Τι απαντήσαμε εμεί για να καταλάβετε σε τι χρησιμεύει ένα συντονιστή η Σαξονία είπε θα ήθελα να γίνει μια μελέτη, αλλά το Ομοσπονδιακό κράτος Γερμανίας δεν θέλει να δώσει ούτε ένα ευρώ. Πλησίασα λοιπόν τους Τσέχους και είπαν ναι συμφωνούμε για να συγχρηματοδοτήσουμε αλλά όχι πλήρως. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το έργο το οποίο τελικά θα κοστίσει αρκετά. Και αρχίσαμε να κάνουμε το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κράτος να αντιλαμβάνεται ότι ακόμη και αν δεν το κάνει αμέσως, πρέπει να κάνει τις μελέτες αυτές παρότι δεν τις χρηματοδοτεί, αλλά ανακαταλάβει ότι και θα πρέπει να συνεργαστούν η Σαξονία, το Ομοσπονδιακό Κράτο, η Τσεχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει για την πρόθεση αυτού του έργου. Τώρα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. οι Γερμανοί έχουν δύο σενάρια. Η πρώτη το πρώτο λέει δεν θα κάνουμε τίποτα διότι αύριο θα φτιάξουμε μια γραμμή υψηλή ταχύτητα. Είναι ένα τρόπο να μην κάνει κανεί τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν, ε, και δεν έχω χάσει κάθε ελπίδα, να γίνουν εργασίες τουλάχιστον μετριοπαθής αλλά αναβάθμισης τη Νιρεμβέργης Σέντιγκ μέχρι τα σύνορα κύριε Κράμερ και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τις μελέτες αρχικά. Όσον αφορά το κομμάτι από το Λίντς προς την Πράγα. Η απαντήση. Το ερώτημα είναι απλό. Και τα δύο κρατή μέλη λένε είναι μια καλή γραμμή, αλλά είναι πολύ ακριβή η συμμόρφωσή τη με τα πρότυπα του έργου προτεραιότητας 22, δηλαδή το να κάνουμε μια δεύτερη γραμμή για να ανέβει στα 140 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι χρήσιμο. Γι' αυτό το λόγο την αφαιρέσαμε από το διάδρομο. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε, είναι ότι και τα δύο κράτη-μέλη μας είπαν ότι αυτή η γραμμή θα έχει τακτική ε, κίνηση, θα ανέβουμε ίσως στα 90 χιλιόμετρα, σήμερα κινείται στα 70, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία της. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει διπλή γραμμή. Μπορούμε λοιπόν να τη βγάλουμε από το έργο προτεραιότητας 22 και να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλους άξονες. Είναι μια συνένεση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων των κρατών μελών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε μάχη γι' αυτό και οι δύο πλευρέ πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διατηρηθεί αυτή η γραμμή. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική της Αυστρίας, την ε, γνωρίζετε και θεωρώ ότι είναι πολύ λογική. βασίστε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης, δηλαδή στο να γίνει η Βιέννη ένα σταυροδρόμι βορανότου Ανατολής Δύσης. Είναι λίγο πιο πέρα από εσά από το Ινσμπρουκ, αλλά σίγουρα απασχολεί ιδιαίτερα τις εθνικές αρχές. Σας το λέω, ε. Τώρα περνάει και από τον Κράτς, μάλιστα, προς το Κόπερ, μετά και να ανοίξουμε και την τεργέστη ώστε να υπάρχει μια διέξοδο ε, προνομιακή προ τη Μεσόγειο από τη Βαλτική μέσω τη Πολωνία και το Κόπερ και το γκράτ ε, προ τη Μεσόγειο. Αυτή είναι η στρατηγική στρατηγική επικεντρωμένη στην σταθμό της Βιέννη, υπάρχει και το Μπρένερ, αλλά αυτά ακούμε στα διαφορά γραφεία, υπουργικά γραφεία, όταν οι υπουργοί μας εξηγούν τις στρατηγικές. Όσον αφορά τώρα τη συντονιστική πλατφόρμα, έτσι την ονομάζω τώρα, όπως έλεγα, είχε μία πολύ απλή διάταξη. 30-40 τόμων, σύνθεση μάλλον, κρατάνε μισές μέρες, επισκεπτόμαστε διάφορα έργα, λειτουργούν όλα πολύ καλά. Ταυτόχρονα, πολύ ειλικρινά, διατηρεί έναν όλο και πιο στενό διάλογο μεταξύ κρατών μελών. Πολύ χρήσιμο και θα καταλήξουμε πιστεύω σε καλύτερο συντονισμό, ειδικά των επενδύσεων στα διασυνοριακά και Λειτουργεί εξαιρετικά από αυτή την άποψη. Ωστόσο και για εμάς είναι εξαιρετικά αποφελές διότι παρεμβαίνουμε τρεις γενικές διευθύνσεις. Αν ήταν μόνο η Γενική Διεύθυνση MOVE θα είχε τις πολιτικές μεταφορών αλλά δεν έχει τις πιστώσεις για τις μεταφορές. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης ταυτόχρονα ώστε να συμπληρώνει η μία το έργο τη άλλη. Δεν μιλάμε απλά για συντονισμό δηλαδή των κρατών μελών. Μιλάμε και για συντονισμό των διαφορετικών δικών μα μέσων. Είναι σταθερός λοιπόν τώρα ο διάλογος, είναι τακτικός και επιτρέπει πολύ σαφώς όταν τίθεται ένα πρόβλημα από ένα κράτος μέλος να το απαντάμε. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αμέσως δίνεται η απάντηση. Τώρα, για να σας μιλήσω για διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το μέσο. Για ποιο λόγο, διότι επιτρέπει να δίνονται κονδύλια για τη συνοχή στην πολιτική μεταφορών. Δηλαδή επιτρέπει να αποφεύγουμε... Ε, εσείς οι ίδιοι λέτε πρέπει να αναπτύξουμε τους σιδηροδρόμους και με τα χρήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο κάνουμε δρόμους, διότι υπάρχουν επιχορηγήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Αντιθέτως θα πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες των κρατών διοικητικέ και τεχνικέ να ανταποκρίνονται σε ε, προσκλήσει ε, υποβολή προσφορών. Δεν έχουν τη δυνατότητα όλα τα κράτη τη Ανατολή. Τώρα η γέφυρα πάνω από το Δούναβι. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τι οδικέ υποδομές κύριε Κράμερ. Αντιθέτω, υπάρχει ένα θέμα που δεν αναφέρατε αυτή τη φορά, να το βλέπετε εδώ. Είναι λίγο χαοτικό βέβαια, αλλά είναι η... ο ποδηλατόδρομος. Ε, θα τη φτιάξουμε. Μπορούμε να προτείνουμε τόσο μαχητικό σας θα να ονομαστεί και Μάικλ Κράμερ. Έτσι, ένας ποδηλατόδρομος πάνω στη γέφυρα του Δούναβη θα μπορούν να κάνουν και ποδήλατο. Όσοι θέλουν αυτά είχα να σας πω τη συνάδελφη για το έργο προτεραιότητας αριθμό 22. Αν και ο σταθμός του Μπριν ε, δεν εντάσσεται στο έργο προτεραιότητας 22, όχι άμεσα τουλάχιστον. Ωστόσο, οι τσεχικές ε, αρχέ δεν μου μίλησαν ποτέ για αυτό το έργο. Είναι πολύ απλό, δεν το έχουν αναφέρει ποτέ το σταθμό του Μπρουνού. Ποτέ δεν ζήτησαν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια από το συντονιστή Ακόμη και ο σταθμό τη Βιέννης ελάχιστα χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκέ πιστώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο σταθμό του Μπρνό αυτή τη στιγμή οι τσεχικέ αρχέ έχουν εκφράσει μόνο δύο ανησυχίε. Τη σύνδεση με τη Γερμανία, τις δύο σύνδεσεις με τη Γερμανία, με την Ερεμβέργη και με τη Δρέσδη. Για να, έχετε μια, να σας δώσω μια πολύ ακριβή εικόνα των ζητημάτων με τα οποία με απασχόλησαν. Ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώνουμε τους πέντε συντονιστές, τους κυρίους Μπάλατς, Μπρίνκος, Κόξ, Σέτσι και Σαβαρή. Τους ευχαριστώ για τις εισηγήσεις τους και συνεχίζουμε με το τελευταίο θέμα και ζητώ συγγνώμη από τον Ρόμπερτ Ζήλε γιατί έχουμε αργήσει μισή ώρα παρόλο ότι προσπάθησα αλλά απέτυχα να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα είναι το θέμα των αερομεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό το, η συμφωνία υπεγράφει τον Ιούνιο μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία για την αεροπλοή, για τις αερομεταφορές και ξεπερνά τις διμερείς συμφωνίες για τις αερομεταφορές μεταξύ μεμονωμένων κρατών μαλών και της Μολδαβίας. Προβλέπει το άνοιγμα των αγορών όσον αφορά την πρόσβαση σε αερογραμμές και αύξηση του δυναμικού σε αμοιβαία βάση. Με τη συμφωνία αυτή, η Μολδαβία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει μια κοινή ε, ε, πολιτική ε, αερομεταφορών και κοινούς κανόνας σε τομείς κλειδιά. Επίσης θα εναρμονίσει την νομοθεσία της η Μολδαβία όσον αφορά τα πρότυπα της περιβαλλοντικής πολιτικής και όλων των άλλων συναφών πολιτικών. Ως αποτέλεσμα η Ένωση και η, Μολδο... η... αερομεταφορή της Μολδαβίας, η αεροπορική εταιρεία θα μπορεί επί αμοιβαίας βάσης να εκτελεί κατευθείαν πτήσεις μεταξύ Μολδαβίας και οπουδήποτε άλλων ε, αερολιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης προβλέπει μια, ε, ένα πλαίσιο επίλυσης ε, των των επιχειρησιακών εμποδίων. Άμεσες και απευθείας πτήσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν με 11 κράτη-μέλη, μεταξύ Μολδαβίας και 11 κρατών μελών. Ε, εγώ προτείνω στην Επιτροπή να επικυρώσει την συμφωνία αυτή αλλά ε, δυστυχώς θα πρέπει η διαδικασία συνένεσης του Κοινοβουλίου να ανασταλεί δεδομένου ότι προέκυψαν διαφορές από το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό το σχέδιο απόφασης ξέπερνα τις αρμοδιότητες των συνθήκων και πρέπει να διορθωθεί. Προβλήματα τέτοιου είδους είχαν προκύψει και στην αρχή αυτού του έτους μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αερομεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Ισλανδίας και Νορβηγίας και ως αποτέλεσμα η Κομισιόν έχει αναλάβει ε, μέτρα κατά του Συμβουλίου τα οποία έχουν ως στόχο την ακύρωση αυτής της απόφασης ε, και το Κοινοβούλιο παρενέβη προς στήριξη της. Ε, από ό,τι ξέρω θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να περιμένουμε για την απόφαση του δικαστηρίου πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση ε, για να δώσουμε τη συνένεσή μας στην ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας από πλευράς Κοινοβουλίου, διότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας και στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας, δεδομένου ότι η προσωρινή εφαρμογή ήδη έχει τεθεί ενισχύ κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πρόεδρος, μάλιστα, λοιπόν, αναστολή και περιμένουμε όλα στάσιμα αυτή τη στιγμή για να δούμε τι θα γίνει τελικά με το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Ο κύριος Κούν θα ήθελα να δικαιολογήσω την αποσία του κυρίου Μαρινέσκου διότι λείπει λόγω των εκλογών στη Ρουμανία. Αλλά θέλω να εκφράσω τις απόψεις του κυρίου Μαρινέσκου. Ε, μου το ζήτησε λόγω της αποσίας του η συμφωνία θα οδηγήσει στο άνοιγμα της αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση, το δυναμικό ε, επί αμοιβαίας βάσεως και θα διαμορφώσει ένα, ένα λεπτό διακόπτη, διακόπτη ο πρόεδρος. Εκτιμώ ιδιαίτερα που εκφράζεται τις απόψεις του κυρίου Μαρινέσκο, αλλά δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτά τα οποία είπε ήδη ο κύριος Ζήλερ. Ε, συμπεράνεται λοιπόν. Ο κύριο Κούν. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι συμφωνούμε με όσα λέει ο κύριο Ζήλε. Συμφωνεί ο κύριος Μαρινέσκου. Ε, και ότι οπωσδήποτε χρειάζεται αυτή η πολιτική και η συμφωνία για τους ανοιχτούς εθέρες θα ήθελα να πω, λέει η κυρία Μάσνα, μην ξεχνάτε το άνοιγμα, τους ανοιχτούς ευρωπαϊκούς ΕΣΕΡΕΣ και ουρανούς κλπ. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία και μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών γυτνίασης. Η κυρία Λίχτεμπερκερ έπρεπε να φύγει και εγώ πολύ σύντομα θα πω ότι συμφωνούμε. Ο κύριος Μπουργκέλ, ε, ελπίζω και εσείς να έχετε την ίδια προσέγγιση. Πράγματι, πρόεδρε, θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω τον κύριο Ζήλε για την εκθεσή του. Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική επειδή επιτρέπει να συμπληρώσουμε αυτό που οικοδομούμε προοδευτικά με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου, δηλαδή έναν κοινό, ένα αέριο χώρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γείτονες χώρες της, όπως υπογράμμισε ο κ. Ζηλέ. Αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, απελευθέρωση των αεροπορικών υπηρεσιών αλλά και βελτίωση των συνθήκων υπό τις οποίες οι ευρωπαϊκές, οι μολδαβικές εταιρείες λειτουργούν σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Μια πολύ ικανοποιητική συμφωνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεση του κύριε Συγητή εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο. Τον συγχαίρομαι λοιπόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν και για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την προσφυγή της Κομισιόν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά του Συμβουλίου. Για να διευκρινίσω ένα πράγμα, σε, κανένα, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πρόβλημα επί του περιεχομένου της συμφωνίας, αλλά θεσμικού χαρακτήρα πρόβλημα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η απόφαση του Συμβουλίου που είναι απόφαση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σε σχέση με την υπογραφή και τη σύναψη της σύμβασης, της συμφωνίας, παραβιάζει τη συνθήκη. Η συνθήκη λέει κάτι απλό, το Συμβούλιο μόνο του εγκρίνει την υπογραφή και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προσφύγει στο δικαστήριο ώστε να θέσει τέλος σε μια κακή συνήθεια, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από θεσμική άποψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και εγώ. Τίποτα άλλο Ρόμπερτ να προσθέσει. Όχι, λέει ο ομιλητή. Σα ευχαριστώ όλου, ο κύριο Ζήλε. σα ευχαριστώ όλου για την κατανόησή σα. Ο πρόεδρος, δεν έχω τίποτα στα διάφορα, απλώς θα σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες 3 ώρα. Το απόγευμα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για την εργασία τους. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, λήξη της συνεδρίασης.